Yeah, yeah, okay. Yeah. Good. So let's try to speak in time for the hearing. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, my... Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κηρύσω την επανέναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί να συζητάμε για τα θέματα του TTIP. για την Συμφωνία Διατλαντικής Συντερικής Σχέσης Εμπορία και Επενδύσεων. Φαίνεται την ημέρα γιατί εκεί και αφιερωμένη στο θέμα του TTIP. Σήμερα θα έχουμε το απόγευμα λοιπόν θα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε με την Επίτροπο Μάλμστρομ για θέματα του TTIP και ιδιαίτερως ε, για θέματα ISDS, θέματα που αφορούν την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτου. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και πώς επηρεάζει τους πολίτες ε, η συμφωνία TTIP. Τα θέματα ISDS είναι από τα πλέον αμφιλεγόμενα τα οποία συζητιούνται στο πλαίσιο της διατραδικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων Και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησαν άλλωστε και διαβουλεύσεις ε, στα σκόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ISDS. Ήταν πολύ άριθμες οι παρεμβάσεις και οι παρατηρήσεις των κρατών μελών για τον πρώτο γύρο των, των διαβουλεύσεων. Η Επίτροπος Μάλμστρομ παρουσίασε και τα πορίσματα, εντόπισε κάποιες προβληματικές ζώνες. Αυτές οι προβληματικές ζώνες ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι επικαλύπτονται με το ψήφισμα του 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσα είχε εντοπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε. Αυτά τα ζητήματα θα εξετάσουμε. Τι θα κάνουμε στο μέλλον σε θέματα προστασίας των επενδυτών και ποιο εργαλείο είναι το πλέον κατάλληλο. Χαίρομαι λοιπόν. Ιδιαίτερος ε, κύριε Επίτροπε που σας έχουμε και πάλι μαζί μας σήμερα. προκειμένου να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί βουλευτές, ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και πάλι. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα δούμε πώς οι επενδύσεις διαμορφώνονται στην διατλαντική εταιρική επενδυτική σχέση. Νομίζω ότι όλα τα ζητήματα, από όλα τα ζητήματα του TTIP αυτό έχει λάβει τη μεγαλύτερη προσοχή έχει προσελκύσει μάλλον τη μεγαλύτερη προσοχή ως τώρα. Δεν είναι περίεργο για τα τελευταία 60 χρόνια οι εθνικές κυβερνήσει των ε, ευρωπαϊκών κρατών διαπραγματεύτηκαν 1.400 διμερείς διαπραγματεύσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Και βεβαίω αυτού του είδου οι τεράστιε επενδύσει έχουν κάνει την Ευρώπη πρωταγωνιστή στην οικονομία, την παγκόσμια για, πολλούς, για πολλέ δεκαετίε. Και έτσι υπήρχε και ζωή κεφαλαίου και δημιουργήθηκαν και θέσει απασχόληση. Από την άλλη, επίση δεν είναι περίεργο που ανησυχούν οι πολίτε, διότι το πλαίσιο για τι διεθνεί επενδυτικέ συμφωνίε έχει αλλάξει εν μέρη εν μέρη λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές ε, εθνικές κυβερνήσεις πλέον είναι από κοινού υπεύθυνε για τις ε, πολυμερείς συμφωνίες. Αυτό προκαλεί περισσότερες συζητήσεις και επίσης με την εμβάθυνση των ε, ε, σχέσεων και των οικονομικών δεσμών η επίλυση διαφορών έχει αλλάξει. Στις διαφορές και στην επίλυση διαφορών μέχρι τώρα είχαμε σαφείς υποθέσεις επενδύσεων. Οι εταιρείε όμως έχουν αρχίσει να πιέζουν τα όρια της ερμηνείας και αυτό έχει οδηγήσει σε καταστάσεις που εκπλήσουν πολλούς. Βεβαίω, βλέπουμε ότι η πραγματικότητα είναι λιγότερο δραματική από ό,τι αρχικά παρουσιάζεται. Οι πλέον αμφιλεγόμενε υποθέσει δεν έχουν εκδικαστεί. Γενικώ, οι επενδυτέ χάνουν τι περισσότερε υποθέσει από ό,τι κερδίζουν και σε πολλέ περιπτώσει πολλέ από τι ε, υποθέσει και τι προσφυγέ του απορρίπτονται. Όμως ε, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα τις επενδυτικές συμφωνίες ε, του παρελθόντος. Επηρεάζουν περισσότερο τους επενδυτές για την ώρα παρά το δικαίωμα των κρατών να ρυθμίζουν. Απλώς το θέμα έχει γίνει καυτό στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο εντατική αυτή η συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πέρσι δημόσιες διαβουλεύσεις για την προσέγγιση μας στην προστασία των επενδύσεων. Ζητήσαμε λεπτομερή ανάλυση αυτού του αποτελέσματος τον Ιανουάριο και σας την παρουσιάσαμε τότε, οπότε δεν θα τα ξαναπούμε. Απλώς η μεγαλύτερη, η πλειοψηφία ε, των ερωτηθέντων ε, απέρριψαν και το TTIP και το ISDS ειδικότερα. Από τις ομάδες ε, των ενδιαφερομένων που είχαμε μεγάλη ποικιλία στην εκπροσώπηση, είχαμε και πολύ διαφορετικές απαντήσεις. Οι διαβουλεύσει βεβαίω δεν ήταν δημοψήφισμα και έδειξαν σαφώ ότι υπάρχει φοβερή επιφυλακτικότητα και ανησυχίε για το σύστημα. Όμως είχαμε και κάποιες πρώτες ιδέες για το πώς να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ε, με μεγάλη χαρά πρέπει να πω ότι και εγώ και ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, ακούσαμε με προσοχή τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Εφόσον έχουμε την αρμοδιότητα για τις επενδύσεις, τα πράγματα είναι σαφή. Το σημερινό πλαίσιο για τις συμφωνίες δεν αρμόζει στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Θέλουμε το κράτος του δικαίου και όχι το κράτος, την επικράτηση των δικηγόρων. Πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις επενδύσεις σε επίπεδο, αλλά πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο καιρό άρχισε να αλλάζει την ε, ε, ε, λειτουργία του ISDS στην συμφωνία με τον Καναδά λόγω χάρη. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω ένα τελικό σχέδιο, απλώς θέλω να σας ακούσω και να δω τις πρώτες σας ιδέες και πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε. να ξεκινήσω δηλώνοντας ίσως το προφανές η αποτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε κανόνε για την προστασία των επενδύσεων και το ISDS μέσα στο TTIP, μέσα στη συμφωνία TTIP. Ξέρω ότι κάποιοι βουλευτέ εδώ έχουν διαφορετική άποψη για διαφορετικού λόγου, αλλά επιτρέψτε μου να σα πω γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Πρώτον, διότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να ε, λυθούν σε σχέση μα με τι ΗΠΑ. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν στι ΗΠΑ και ήδη το σύστημα πύληση διαφορών του είναι εύρυθμο. Τι να μας ανησυχεί. Αληθεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα τέτοιο σύστημα δικαστικό που είναι πολύ καλής λειτουργίας η διακριτική μεταχείριση ή άλλα τύπου προβλήματα είναι πολύ μικρότερα από ό,τι στο υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση για του ξένου επενδυτέ. Η ε, συμπερίληψη επένδυση των επενδύσεων σε αυτή τη συμφωνία θα κάλυπτε το χάσμα. Το ISDS είναι ω μηχανισμό ο μόνο τρόπο να επιβάλλουμε αυτή την επίλυση. Ε, διότι το εθνικό δίκαιο για την ώρα δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανεί στα αμερικανικά δικαστήρια. Ο μηχανισμό θα ε, μπορούσε να εμποδίσει τι μικρέ εταιρείε από την πρόσβαση στο σύστημα. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μικρό ο αριθμό των υποθέσεων που ε, εκδικάζονται, κυρίω για τι μεγάλε εταιρείε, όπω γίνεται τώρα και στον ΠΟΕ. Και η Ευρώπη θα ήταν σε μειονεκτούσα θέση σε σχέση με, την, ε, με τι Ηνωμένε Πολιτείε, κάτι που συμβαίνει ήδη με, την, ε, με τον Καναδά ή την Ιαπωνία, λένε κάποιοι. Και επίση, εννέα έχουν ήδη συμφωνίε που ε, ισχύουν στη σχέση του με τι Ηνωμένε Πολιτείε, και αυτό δεν τι εμποδίζει να εφαρμόζουν το σύνολο του κεκτημένου από το 2004. Όμω είναι προβληματικό διότι δεν έχουν συμπεριλάβει τι μεταρρυθμίσει που εγώ θεωρώ απαραίτητε για να επανασορροπηθεί το σύστημα ε, υπέρ τη ε, σωστή διεξαγωγή τη διαδικασία. Με του κανόνε του TTIP κάποιοι λένε ότι είναι ε, και ότι θα ισχύσει το γνωστό σύστημα επίλυση διαφορών. Κατά τρίτον, οι ΗΠΑ είναι το αναγκαίο σημείο αφετηρία για την αναθεώρηση το 3.000 επενδυτικών συμφωνών που υπάρχουν σήμερα ανά τον κόσμο. Εμεί έχουμε τη μερίδα του λέοντο από, την, ε, από τις υπάρχουσες ε, συμφωνίες με, την άμεση, με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Άλλωστε, οι, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμερίζονται την ε, μεριμνά μα για την προστασία του δικαιώματος προσφυγής. Αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο αφετηρία λοιπόν για να αναθεωρήσουμε τι 1.400 συμφωνίε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλου εταίρου, μεταξύ των οποίων και είναι εξελίξει και Μεταξύ αυτών ο Καναδά διαφέρει όμω συμφωνία αυτή έχει διπερατωθεί και έχει ήδη ενσωματώσει πολλέ από τι καλέ ιδέε που έρχονται από του βουλευτέ. Ε, Ε, για πρώτη φορά υπάρχει μνήμα στο δικαίωμα ρύθμιση. Με την καλύτερη διευκρίνηση του δικαιώματο αυτού και την ισότιμη μεταχείριση αλλά και την ε, έμεση ε, απαλωτρίωση, να προστατεύουμε τα δικαιώματα των κυβερνήσεων ε, και των διαιτητών για το πώ θα ερμηνεύσουν του κανόνε. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδά δεν συμφωνήσουν με την απόφαση ενό διαιτητή, μπορούν να ε, εκδώσουν μια μονομερή δήλωση για το πώ θέλουν να γίνει η ερμηνεία. Άλλωστε, σε αυτή τη συμφωνία για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε και ένα κώδικα συμπεριφορά για του διαιτητέ. Και ανοίξαμε την πόρτα για ένα μηχανισμό επίλυση για το μέλλον. Έτσι υπάρχουν απαιτήσει διαφάνεια για την διεξαγωγή ε, ε, εκδίκαση των υποθέσεων και ε, θα πρέπει οι προσφεύγοντε να εγκαταλείψουν την εκδίκαση σε εθνικά δικαστήρια εφόσον θέλουν να έχουν προσφυγή στο μηχανισμό. Θα πρέπει να δούμε συλλογικά τι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο TTIP και ε, πετυχαίνοντα τη συμφωνία και τη καναδική κυβέρνηση. Δεν θέλω όμω εδώ να σα δώσω ελπίδε, διότι από την προοπτική του Καναδά η συμφωνία αυτή έχει περατωθεί, έχει ολοκληρωθεί και έχει τελειώσει. Επιπλέον, τα οικονομικά ε, συμφέροντα, τα οικονομικά ωφέλη που έχουμε αποκύψει από την συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά είναι ήδη πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο Καναδά δεν θα θελήσει να ανοίξει άμεσα νέα κεφάλαια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άλλωστε, υπάρχουν ρήτρε αναθεώρηση από τη συμφωνία που θα μα επιτρέψουν να τα ξαναδούμε αυτά στο μέλλον και ο Καναδά συμμερίζεται τι απόψει μα για, για τη σημασία του δικαιώματο του ρυθμίζει. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν, νομίζω ότι τα θέματα του να περιλάβουμε τι επενδύσει στο TTIP δεν αφορούν το κατά πόσον ε, θα το κάνουμε ή όχι, αλλά αν μπορούμε να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, αν μπορούμε να έχουμε μια νέα μορφή επίλυση διαφορών που να διατηρεί τι θετικέ συνέπειε και επιπτώσει και όχι τι αρνητικέ. Η απάντηση πιστεύω είναι θετική. Διότι αν πάρουμε τη συμφωνία ε, ΣΕΤΑ, την ε, ει βάθο και ολοκληρωμένη οικονομική, συμφωνία οικονομική συνεργασία, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με, ένα καλό, με μια καλή αφετηρία. Βέβαια αυτό είναι η αρχή της συζήτησης και όχι ολοκλήρωση της. Όμως το βασικότερο θέμα που έχει εκφραστεί από τους περισσότερους που ανησυχούν είναι ότι η επίλυση διαφορών για τις επενδύσεις στο TTIP θα είναι ένας φραγμός για την ευγενή μας παράδοση της υψηλής ε, ρύθμισης. Ε, θα υπάρχει πολύ περιθώριο για να... Ε, αμφισβητήσουν του κανόνε και τι νομοθεσίε οι επενδυτέ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προστατεύσουμε τι δραστηριότητε των επενδυτών, λένε κάποιοι άλλοι. Αυτέ είναι οι σημαντικέ μερίμνε τι οποίε θα πρέπει να τι καλύψουμε στο νέο επενδυτικό σύστημα επίλυση διαφορών. Αυτό πιστεύω να μπορεί να γίνει με δύο τρόπου. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει ένα σαφέ άρθρο στο κείμενο που να ορίζει ότι οι κυβερνήσει μπορούν να συνεχίσουν τι δημόσιε πολιτικέ και του στόχου του και το επίπεδο προστασία που θεωρούν κατάλληλο και δέον. Μια άλλη πιθανή αλλαγή θα έπρεπε να ασχοληθεί με τα επιχειρήματα που λένε ότι οι επενδύτες μπορούν απλώς να μηνύσουν διότι αλλάζει το ρυθμιστικό περιβάλλον. Δηλαδή ότι οι επενδυτέ θέλουν ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και ότι έτσι θα ανοίξει πόρτα σε υποθέσει που απλώ θα έχουν ω αφορμή την αλλαγή τη νομοθεσία. Η δική μα άποψη είναι ότι οι κανόνε προστασία των επενδύσεων δεν προσφέρουν καμία εγγύηση για του επενδυτέ ότι το νομικό καθεστώ εντό του οποίου επένδυσαν στην αρχή θα παραμένει διαρκώ το ίδιο. Εκτό από κάποιε βασικέ βεβαίω ε, ρήτρε προστασία. Ε, λόγω χάρη τα δικαιώματα ιδιοκτησία ε, και πνευματική ιδιοκτησία. Ο δεύτερο τρόπο αφορά το πώ ε, λειτουργούν τα δικαστήρια. Πολλοί ανησυχούν ότι δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων με το σύστημα, διότι οι διαιτητέ είναι και δικηγόροι και μπορεί να επηρεάζονται επιχειρηματικά από του επενδυτέ στο μέλλον. Η δική μα άποψη εδώ είναι ότι οι κυβερνήσει, πολύ πριν ε, εκδικαστούν ε, οποιασδήποτε υποθέσει, θα πρέπει να διορίσουν έναν κλειστό κατάλογο αξιόπιστων διαιτητών που θα αποφασίσουν για τις υποθέσεις του TTIP. Ε, και θα πρέπει ε, αυτοί να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Λόγω χάρη να, είναι, ε, να μπορούν να έχουν τις ικανότητες να είναι δικαστές βάσει του εθνικού του συστήματος. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα μόνιμο δικαστήριο για τις επενδύσεις με μόνιμους δικαστές που δεν θα επηρεάζεται τις μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Κάποιοι λένε ότι η καλύτερη ιδέα είναι αυτή ένα μόνιμο, ένα επίσημο δικαστήριο. Και εγώ το θεωρώ πολύ καλή ιδέα. Ήδη μου το σκέφτονται και θέλουν να διαμορφώσουν μια σχετική πρόταση. Χρειαζόμαστε ωστόσο ένα δικαστήριο που θα ξεπερνά τα όρια του TTIP. Δηλαδή ένα δικαστήριο για πολυμερεί υποθέσει που θα κάνει μια καλύτερη χρήση των πόρων και που θα έχει περισσότερη νομιμότητα. Ε, αυτό θα είναι ένα μέσο πρόθεσμο στόχο, τον οποίο πρέπει να επιδιώξουμε μαζί με τι ε, διαπραγματεύσει μα με τι ΗΠΑ. Ελπίζω να κερδίσω τη στήριξη του Κοινοβουλίου εδώ και να μου πείτε κι εσεί πώ θέλετε να προχωρήσουμε. Τρίτον, οι προσφυγέ και οι εθέσει. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα ε, ε, ε, έφεσης, υποβολής έφεσης στο σύστημα ASDS και στο TTIP είναι κάτι που πρέπει να το λύσουμε. Θα ήταν καλό να υπάρχει ένα τέτοιο εφετείο με μόνιμα μέλη και πάλι εντός της συμφωνίας TTIP. Θα υπάρχει έτσι συνέπεια στην ε, ε, ερμηνεία και την αναθεώρηση των αποφάσεων. Επίση, ένα μηχανισμό προκολή έθεση για του άλλου ε, πολιτικού εταίρου και όσου διαπραγματευόμαστε, όπω ο Καναδά. Ένα τέτοιο εφετείο θα μα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε έναν σταθερό μηχανισμό πολυμερή για την υποβολή εφέσεων. Και μετά πρέπει να δούμε το θέμα της σχέσης μεταξύ του εγχώριου νομικού συστήματος και του ISDS, διότι το εσωτερικό μας νομικό σύστημα θα πρέπει να είναι αυτό που ε, θα πετανεύει, θα βρισκεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν είναι το ISDS άδικο, δηλαδή λένε κάποιοι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να ε, ανακαλέσουν, να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων οι επενδυτές. Οι επενδυτές θα πρέπει να επιλέξουν από την αρχή όμως μεταξύ εθνικού δικαστηρίου ή του μηχανισμού ISDS. Δεν θα επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν το ISDS εφόσον η υπόθεσή του έχει εκδικαστεί σε εθνικό δικαστήριο. Ωστόσο, η αρνητική συνέπεια από κάτι τέτοιο θα ήταν δυστυχώ να ενθαρρύνουν τι εταιρείε πάντοτε να αποφεύγουν τα εθνικά δικαστήρια και να τα παρακάμπτουν. Μια δεύτερη επιλογή, και εδώ θα ήθελα να ακούσω τι απόψει σα, είναι ίσω να φροντίσουμε οι επενδυτέ να αποφύγουν, να καταλήψουν οποιαδήποτε ε, προσφυγή έχουν ε, ε, ξεκινήσει εφόσον προσφύγουν στο ISDS. Δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνει προσφυγή στο SDS εφόσον ο επενδυτή έχει αποφασίσει να ε, ε, εξαντλήσει τα ε, εγχώρια ένδικα μέσα. Δεν μπορεί να γίνει τέτοιο άλμα, τέτοια παράκαμψη. Αυτέ είναι οι ιδέε που έχουμε για την ώρα, είναι προκατακτικέ μα ιδέε, το τονίζω και θέλουμε να τι συζητήσουμε μαζί σα. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, για να ακούσω τι δικέ σα τι απόψει και τι συμβουλέ. Και την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει, μια, ε, υπάρχει ένα τύπο Υπουργικό Συμβούλιο ε, στη Ρήγα. Θα συζητήσω εκεί και με του Υπουργού Δικαιοσύνη και κατόπιν αυτών ελπίζω να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα την Άνοιξη, ώστε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι μια σοβαρή ε, προσπάθεια να φωτίσουμε αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα και ε, περιμένω την οπικοδομητική μας συζήτηση με εσά για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Με αυτήν την κάπως μακρά εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν σημαντικό λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος. Ε, υπομονώ για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και στους κοιότητες εισηγητές. Καταρχάς, για να απαντήσουν στις ε, παρατηρήσεις ε, της ε, Επιτρόπου. Εισηγητής, όπως γνωρίζετε, είμαι εγώ, άρα θα μιλήσω με την ιδιότητα του εισηγητή τώρα. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις, κυρία Επιτροπέ. Καταρχάς, για το ερώτημα του ποιο εργαλείο χρειάζεται για την προστασία των επενδύσεων στη τελική ανάλυση. Το ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για μια προστασία των επενδυτών είναι θεωρώ ανδιαμφισβητητό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ίση αντιμετώπιση δαπών και είμαι ε, επενδυτών. Να μην υπάρχουν ούτε πλέον εκτήματα αλλά όχι και, και μειονεκτήματα. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί την αρχή που θα διαμορφώσει τη σύμβαση και στη συνέχεια θα κληθούμε να αποφασίσουμε και να συζητήσουμε ποιο είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο προς το σκοπό αυτό. Το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο κατέρτισα αναφέρει σαφώς την απόψή μου ότι αυτή η αρχή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν θα να, δεν χρειαζόμαστε καμία εξοδικαστική αρχή γιατί η ιστορία έχει καταδείξει ότι δεν υπάρχει σημαντική διακριτική μεταχείριση υπέρ ή κατά κάποιων επενδυτών. Από πλευράς οικονομικής δηλαδή δεν υπάρχει η ανάγκη αυτή. Και κατά το δεύτερον, το εργαλείο αυτό θα προκαλούσε πολλά πολιτικά ζητήματα, πολιτικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αυτή η θέση παραμένει για να προστατεύσουμε την αρχή αυτή. Θα πρέπει να δούμε ποιος θα εισαγάγει και πότε τέτοια συστήματα. Με τη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, έχει ήδη καταρτιστεί συμφωνία και εκ των εκ των υστέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το σύστημα αυτό ή για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις ε, με τον Καναδά. Το εργαλείο αυτό δεν εισήχθη από τον Καναδά. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε πότε χρειαζόμαστε τα εργαλεία αυτά για να εγγυηθούμε την αρχή αυτή της αντιμετώπισης των επενδυτών. Μια δεύτερη παρατηρήσει, κυρία Επιτροπέ. Είπατε ότι ο Καναδάς και η συμφωνία σχετική έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε φυσικά τον ίδιο προβληματισμό και εδώ, σε πολλούς τομείς. Οι ανασφάλειες ε, τις οποίες περιγράψατε, οι αβεβαιότητες που προκύπτουν αναφορικά με το ISDS, ε, μας ταλανίζουν και εκεί. Δεν καταλαβαίνω τη λογική λοιπόν του πώς μπορούμε αφενός να δηλώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με το παλιό ISDS και ως εκ τούτου συζητούμε ένα καινούριο ISDS. Στο ίδιο μορφότυπο όμως με το παλιό και το εξετάζουμε ως σύστημα που θα ενταχθεί σε μια συμφωνία. Θα πρέπει θεωρώ να σκεφτούμε καλύτερα το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη συμφωνία με τον Καναδά. προκειμένου τελικά να μην πληχθεί μια συμφωνία η οποία κατά τα άλλα είναι εν γέννη καλή. Μία τρίτη παρατηρήση. Όντως για τις προτάσεις που κάνατε. Νομίζω ότι αυτά αποτελούν σωστά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ε, κατοχυρώσουμε την αρχή αυτή, όχι όπως στη συμφωνία με τον Καναδά στις θεολογικές σκέψεις, αλλά στο διδακτικό, προκειμένου να υπάρχουν ανεξάρτητοι δικαστές που θα μπορούν να αποφασίζουν αμερόληπτα και ανεξάρτητα. Να υπάρχει ένας κώδικας ε, δεντολογίας, να υπάρχει μια λογική δυνατότητα αναθεώρησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνεται όπως γίνεται σήμερα διπλή χρήση και αξιοποίηση του δικαστικού συστήματος και των εθνικών κανονισμών. Όλα αυτά λοιπόν θα οδηγούσαν στη δημιουργία ενός διεθνούς ε, δικαστηρίου όπου θα μιλάμε πραγματικά για ένα πραγματικό δικαστήριο όχι μόνο για δικαστικές υπηρεσίες όπως προβλέπονται σήμερα από το ISDS αναρωτιέμαι μήπως αυτός θα έπρεπε να είναι ο απότερος στόχος των διαπραγματεύσεων. Να βρεθεί επαρκής αριθμός των κρατών, κρατών που υπό τη σκέπη του ΠΟΕ θα δημιουργούσε, θα εγκαθίδρυε μια τέτοια, ένα τέτοιο διεθνές δικαστήριο. Αυτό ωστόσο σημαίνει παράλληλα ότι αυτό θα έπρεπε να καταστεί αρχή των διαπραγματεύσεων. Να προωθήσουμε δηλαδή την διαιτησία αυτή, όπως προβλέπεται και στο σχετικό άρθρο προστασίας της συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, όπου προβλέπονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις για να βρεθεί ένα κοινό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα υποστήριζα σίγουρα το σημείο αυτό. Αυτά είναι συντομία από δική μου πλευρά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο την κυρία Κουιστχάουτ Ροβόλ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας για πολλωστή φορά εδώ στην Επιτροπή μας και για το γεγονός ότι τόσο ανοιχτά μας παρουσιάζεται πως έχει η κατάσταση. Θα πρέπει να σας πω ότι είμαι θετικά εκπληκτή από τις προτάσεις σας. Πηγαίνουν πολύ μακριά. Και μάλιστα στην κατεύθυνση επί της οποίας έχουμε συμφωνήσει σε διάφορους κύκλους ανεπίσημα Συμφωνώ με την απόψή σας ότι στην προκειμένη περίπτωση ένα, ενός τύπου διακανονισμός διαφωνιών από κράτος σε κράτος δεν θα είχε οποιοδήποτε νόημα. Αντίθετα με τον προηγούμενο μιλητή πρέπει να ομολογήσω ότι και οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις μπορούν να αποφεληθούν από τέτοιες ε, δικαστικές ε, υπηρεσίες, ε, επιδετησίες μάλλον, αρχές επιδετησίες. Στη Γερμανία έχουμε παραδείγματα όπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις δικαιώθηκαν τον τρόπο αυτό. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πολλά σε ό,τι αφορά θέματα τέτοιων συμβάσεων, πολλά εξαρτώνται από τα μόσπονδα κρατήδια και όχι από το μόσπονδο κράτο. Και εδώ φυσικά έχουμε πρόβλημα αν το μόσπονδο κρατήδιο δεν ε, δείξει ενδιαφέρον για όσα έχουν συμφωνηθεί σε διεθνέ επίπεδο. Ποια θα είναι η σχέση λοιπόν. Έστω ότι υπάρχει αυτή η επενδυτική προστασία. Σήμερα το πρωί δήλωσα ότι θα πρέπει να υπάρξει τροποποιημένη προστασία επενδυτών στα πλαίσια μιας διεθνούς σύμβασης. Πώς λοιπόν θα πετύχουμε μια εγγύηση κοιτώντας ε, και την, το τοπικό επίπεδο ότι θα υπάρχει αυτή η προστασία και εφαρμογή. Η μείωση των αγωγών ερμηνεύεται με αρνητικό ή θετικό τρόπο από κάποιους. Αλλά καλό είναι σε κάθε περίπτωση να γνωρίσουμε και να περιγράψουμε το τι μπορεί να αποτελέσει βάση για αγωγή, για καταγγελία. Να υπάρχει κατάλογος για τις, ε, τα δυτικά όργανα, εδώ συμφωνούμε, να υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Και να υπάρχει και δυνατότητα τροποποίησης το θέμα ενός διεθνούς ε, διαιτητικού δικαστηρίου στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ενδεχομένως. Μέσω πρόθεσμα θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυνατότητα. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ας προσπαθήσουμε σε πρώτη φάση να καταθήσουμε ένα ομογενές, διαφανές και συνεκτικό σύστημα. Μια συνεκτική διαδικασία. Να συμφωνήσουμε από αυτού και βάσει της εμπειρίας αυτής να συνεχίσουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, γιατί το τρίτο ζήτημα το οποίο θίξατε για τα θέματα δηλαδή ενστάσεων θα πρέπει και προσφυγών και εφέσεων θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι τελικά ο τελικός αρμόδιος, ποιος θα μπορεί τελικά να λαμβάνει την τελική απόφαση, γιατί θεωρώ ότι ένα από τα δύναμα σημεία είναι το εξής Πώς διαμορφώνεται το σύστημα εφέσεων. Εγώ όταν να σας πω, φυσικός είμαι, μπορώ να κάτσω και να ακούσω ό,τι μου πείτε. Αυτά που θα έχουν να πούνε οι πιο σχετικοί νομικοί. Σχέση προστασίας, επένδυσης σε σχέση με τα εθνικά δικαστηρία. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο και κάποια από τις ε, εναλλακτικέ θα διακριθεί ως πλέον κατάλληλα. Κατάλληλη. Ένα πράγμα όταν έχουμε συζητήσει στις συζητήσεις μας. Λέμε τι, με τι συμφωνούμε, με τι διαφωνούμε. Αλλά υπάρχουν τόσο πολλές διμερείς συμφωνίες. Αν δεν συμφωνήσουμε για μια νέα μορφή επενδυτική προστασία, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διμερεί συμφωνίε. Υπάρχουν εννέα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ασφαλίζονται και προστατεύουν διαφορετικά του επενδυτέ του από τα υπόλοιπα 19. Αυτό σε μια συμφωνία διμερή μεταξύ μεγάλων ομάδων όπως είναι η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το πάρα πολύ περίεργο. Δεύτερο στοιχείο. Θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τι γίνεται με το εξή. Αν συνεχίσουν να ισχύουν όλα αυτά, τι σημαίνει αυτό για τις αμερικανικές επενδύσεις ε, στην Ευρώπη, οι οποίες επίσης θα τυχάνουν διαφορετικής προστασίας ανάλογα με το πού πραγματοποιούνται. Σε ποιο κράτος γίνονται οι επενδύσεις. Τελευταίο σημείο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι έχει διευκρινιστεί, είναι η σχέση ΣΕΤΑ με TTIP. Στο σημείο αυτό. Συχνά αναφέρουμε ότι το ΣΕΤΑ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για το TTIP. Αυτό είναι κάτι πρόσφατο στις τελευταίες συζητήσεις, στους τελευταίους μήνες, στις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα επενδυτική προστασία, αλλά ιδιαίτερα στον τομέα αυτό. Όταν λέμε ότι θέλουμε κάτι σαν το ΣΥΤΑ-ΨΥΝ, δηλαδή, τι εννοούμε, θα κάνουμε μια διαπραγματεύση του συμφωνία ΣΥΤΑ. δηλαδη τι εννοουμε θα κανουμε νέα διαφωνώ με τον ε, προλαλήσαντα. Θεωρώ ότι το πακέτο ΣΕΤΑ είναι ένα πακέτο όπου κάθε πλευρά θα πρέπει να κάνει συμβιβασμού. Αυτό φυσιολογικό είναι σε κάθε είδου διαπραγμάτευση, αλλά αν ανοίξουμε κάτι μόνο μερό σε ένα σημείο, φοβάμαι και προβλέπω ότι και οι Καναδοί που δεν συμφωνούν με όλα τα σημεία και με κάποια σημεία τα οποία πραγματικά θέλαμε να περάσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι και έτσι θα ξανανοίξουν το πακέτο δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί απαραίτητο το σκοπό μας. Ωστόσο, και αυτό πραγματικά είναι η τελευταία παρατηρήση που έχω να κάνω, σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδυτών, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εξέτασης. Ε, μπορεί να κινηθούμε προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να δείξουμε ανοιχτή, ανοιχτό πνεύμα, να ακούσουμε όσο πιο πολλές προτάσεις γίνεται, να ακούσουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατόν, με επίγνωση της κατάστασης να αποφασίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε 11 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο ακόμα. Μέχρι τις 4 έχουμε χρόνο. Και μετά η Επίτροπος θα πρέπει να έχει και την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ως εκ του θα πρότεινα να περιορίσουμε το χρόνο ομιλία σε δύο λεπτά. Έμα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα βάλω τα δυνατά μου και ευχαριστώ την Επίτροπο που ήρθε προκειμένου να βρούμε από κοινού ένα δρόμο να προχωρήσουμε. Γιατί μέχρι στιγμής βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο στο TTIP, αλλά όχι μόνο στο TTIP. Και με τις άλλες συμφωνίες που έχουμε επιτάπητος έχουμε ένα πρόβλημα, ένα διέξοδο. Ακόμη και με τη ΣΕΤΑ πρέπει να το ξεμπλοκάρουμε. Οπότε πρέπει να δούμε τι μορφή πρέπει να πάρει αυτή η επενδυτική προστασία. Γιατί συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μορφή επενδυτική προστασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πιο διεξοδικά τις, προσπά, τις προτάσεις και να δούμε ποιος είναι ο καταλληλότερος μηχανισμός για να προχωρήσουμε και να δώσουμε μορφή στην προστασία των επενδυτών. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει μία νυχτή. Ό,τι και κάνουμε πάντως θα πρέπει να φροντίσουμε να ακολουθήσουμε τη σωστή άγουσα και να είμαστε διαφανείς για να προσετεριστούμε και την κοινή γνώμη. Επίσης, ε, είπαμε ότι θα περισσότερες αντιδικίες θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι τέτοιες μορφές επενδυτικής προστασίας ε, έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Και στηρίζουμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ε, είναι πολύ συσταλτική η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών. Όποιο και μηχανισμό επιλέξουμε, δεν εθαρρύνουμε την αντιδικία. Απλώς θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών για να μπορούν να επενδύουν. Δεν εθαρρύνουμε ε, την ε, δικομανία. Σε καμία περίπτωση. Αυτή λοιπόν είναι η αρχική μου σκέψη και επίσης να φροντίσουμε να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα και να δούμε ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας όλων αυτών των προτάσεων ε, και τι λύση θα βρούμε και για την συνολική συμφωνία, την εμπορική και την οικονομική με τον Καναδά. Τι προτάσεις έχουμε κάνει στους Αμερικανούς και τι δεσμεύσεις έχουμε λάβει από τους Καναδούς στην όλη διαδικασία. Πάντως, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να περάσουμε από μια αρνητικότητα σε μια προσπάθεια ανέβρεσης θετικών λύσεων για να προχωρήσουμε και μάλιστα επικοδομητικά και στις διαπραγματεύσεις με το TTIP και στις άλλες μας εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ, Χέρμαν Σόλτς. Όχι, συγχωρέστε με κύριε Λάντουπερ, δεν ήξερα ότι ε, αντικαθιστάτε την κυρία Σάκε ως κοιόδης. Ε, σας ε, ευχαριστώ. Εμεί οι φιλελεύθεροι έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν καταρχάς κυρία Επιτροπέ που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα γιατί ένα κομμάτι της μεγάλης διαφάνειας της Επιτροπής είναι πραγματικά φανερό και το καλωσορίζουμε. Ένα πράγμα είναι σαφές. Θα γίνει ένα τμήμα τη συζήτηση αυτή το οποίο δεν θα πιστεί. Αρκεί να κοιτάξουμε το Twitter, να δείτε τι γίνεται. Χαμός γίνεται. Να σταματήσουμε το TTIP. Μερικούς δεν θα μπορέσουμε να τους πείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτοί που μπορούν να πιστούν Νομίζω ότι ωφελήθηκαν πάρα πολύ από τις καλές ιδέες που άκουσαν από σας σήμερα. Το να πούμε ότι είτε θα κινηθούμε προς την, επένδυση, την προστασία των επενδυτών, είτε προς την εθνική, ε, εθνικούς κανονισμούς, είναι καλή και θεωρώ ότι η ιδέα να δημιουργηθεί ένας εξάρτητος, ε, μια ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία για την υπηρεσία θα είναι καλή. Το κατά πόσο θα γίνει αυτό για το TTIP είναι άλλο θέμα. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη κατά πόσο θα ήταν εφικτό να υπάρχει ένα μόνιμο τέτοιο δικαστήριο στο οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί και το TTIP. Τελευταίο σημείο. Μου κάνει εντύπωση πάντα το πόσοι βγαίνουν και λένε ότι στη ΣΥΠΑ υπάρχει ένα πολύ καλά λειτουργούν σύστημα, δικαστικό σύστημα. Ναι, όντως πρόκειται για ένα σύστημα δικαστικό το οποίο είναι πολύ λειτουργεί πάρα πολύ καλά, το οποίο αντιμετωπίζουμε εμεί στην Ευρώπη με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό και δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις μα που επενδύουν στη ΣΥΠΑ να πρέπει να εξαρτώνται από τη δικαιοδοσία κάθε πολιτείας, όπου δεν ξέρουν τι διακριτική μεταχείριση θα υποστούν. Μα αυτοί που λένε ότι το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ είναι τόσο φανταστικό είναι οι ίδιοι που επικρίνουν την συμφωνία και λένε δεν θέλουν να είμαστε στο έλεος του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ. Τελευταίο σημείο. Αν υπάρχει αν υπάρξει τελικά η συμφωνία TTIP, αλλά χωρί να συμφωνήσουμε για ένα σύστημα προστασία των επενδυτών και πάλι έχουμε κάποια προστασία των επενδυτών, γιατί υπάρχουν οι διμερεί συμφωνίε. Ο κ. Σόλτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα που μα δίνεται επανειλημμένα να εκφέρουμε γνώμη και να συζητήσουμε για το θέμα τη συμφωνία TTIP και να σα πω ότι είμαι από του επικριτές του ISDS. Το είπα και σήμερα το πρωί. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεση για την Ιταλική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων που προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι θεωρώ ότι το ISDS μπορεί να πάει στα σκουπίδια της ιστορίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την επίλυση διαφορών σε ένα τομέα, ο οποίος, το οποίο πλέον δεν συμβαδίζει και δεν συνάδει με τον 21ο αιώνα. Και γιατί, γιατί είναι σύνθετη η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Ιδιωτικό σύστημα επιδιατησίας σε, για μια συμφωνία διεθνούς δικαίου. Δηλαδή τα κράτη συνάπτουν μια συμφωνία με άλλα κράτη όπου η υπηρετησία ανατίθεται στα χέρια του ιδιωτικού δικαίου. Γιατί στον 21ο αιώνα να γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ εμπιστοσύνη στις ε, μελλοντικέ μορφές επενδυσίας. Γιατί υπάρχει ένα επιχειρηματικό κλίμα, μια επιχειρηματική ατμόσφαιρα σε ό,τι αφορά την επενδυτησία. Για το ποιος μπορεί να υποστηριχθεί ή να κατηγορηθεί και να λειτουργήσει ως κατηγορούμενος ε, ή ως ενάγων σε ποιες περιπτώσεις. Αναγνωρίζω τις απόπειρες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αυτή η κριτική, η οποία συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό, να τη αντιμετωπίσει. Είχε προσπαθήσει να το κάνει και στα πλαίσια τη συμφωνία ΣΕΤΑ αλλά πιστεύω ότι δεν φτάνουν οι προσπάθειες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν ε, απομακρυνόμαστε, δεν καταφέρνουμε να επιλύσουμε την ουσία του θέματος. Χρειαζόμαστε ένα διεθνέ δικαστηρίο το οποίο θα είναι δεσμευτικό για όλα τα μέρη από πλευρά διεθνού δικαίου. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, κοινή λογική. Το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί με τη λογική αυτή κατά το παρελθόν και θα πρέπει να ξεφύγει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, Τζανιζέλο. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Μας εξηγήσετε ότι το σύστημα είναι κάπως τρευλωμένο, κακοφτιαγμένο και ότι θα προσπαθήσετε να το βελτιώσετε. Αλλά δεν μας αποδείξετε προς τι αυτό το σύστημα. Γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα. Γιατί η Ευρώπη, η Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ανάγκη αυτό το σύστημα. Μάλιστα, διαβάζοντας τι μελέτες τη Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΣΑ και την κατάσταση των διατλαντικών επενδύσεων, δεν έχουμε ούτε έναν οικονομολόγο σήμερα που να λέει ότι αυτό το σύστημα προστασίας των επενδύσεων ή των επενδυτών με, ευρω... ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια προστατεύει τις επενδύσεις. Ούτε μια οικονομική μελέτη δεν λέει ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου ιδιωτικού δικαστηρίου διαιτητικού ευνοεί τις επενδύσεις. Ε, μας είπατε ότι έχουμε 1.400 συμφωνίες ε, που περιλαμβάνουν και το ISDS, άρα να το διαιωνίσουμε. Δηλαδή, είναι τόσο θετική η κατάσταση, έχουμε τέτοια ευτυχία στις διεθνείς σχέσεις και τέτοια ευεξία ώστε να επαναλαμβάνουμε τις ρυθμίσεις του παρελθόντος. Γνωρίζετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μέχρι τώρα συστημάτων ε, εφαρμόστηκαν με, υπα... με υπανάπτυξες αναπτυσσόμενες χώρες, με χώρες Ανατολής πριν την ε, προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρήσαμε ότι στις χώρες αυτές δεν υπήρχε ούτε ε, αξιόπιστο νομικό σύστημα, ούτε κράτος δικαίου. Και όταν είπε το πρωί ο κράτος συνάδελφος ότι χρειαζόμαστε το ISDS, γιατί αν θέλουμε αλλοδαπούς επενδυτές θα πρέπει να μπορούμε να τους πούμε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουν να ε, αποταθούν στα δικαστήριά μας, αυτό είναι παταγώδης αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μηχανισμός που τη χάνει προστασίας. Είπατε ότι θα τη το αγρίμι, ε, ότι θα βελτιώσουμε το μηχανισμό. Ο λύκος όμως ε, δεν αλλάζει τη φύση του, ακόμη και αν αλλάξει το τομάρι του. Δεν πρόκειται να βελτιώσουμε το σύστημα. Επίσης, ε, έχουμε τις συμφωνίες Apple Ιρλανδίας και Starbucks Ολλανδίας. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να στυλιτεύσει και να επιβάλλει κυρώσεις αυτές τις φορολογικές συμφωνίες και να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις ε, να καταβάλουν τους φόρους ε, που διέφυγαν. Και φυσικά ε, η Starbucks, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το Δυτικό Δικαστήριο για να αποφύγουν να καταβάλουν τους φόρους που χρωστούν. Τώρα, ψηφιακή οικονομία. Το παρουσιάζουμε ως μείζον επίτευγμα. Και σήμερα 85% ε, ε, των επιχειρήσεων ε, της ψηφικής οικονομίας είναι αμερικανικές. Οι κανόνες του παιχνιδιού χαράζονται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα θέλουμε ψηφιακή οικονομία εδώ, θα πρέπει να χαράζουμε και να μπορούμε να επιβάλλουμε του κανόνε μα. Και με το ISDS αποκλείται να τα καταφέρουμε. Επίση, έχουμε ένα ανώτερο σύστημα, καλύτερο, που μάλιστα με ένα τέτοιο σύστημα θα διακυβεύσουμε, θα υπονομεύσουμε τα εσωτερικά μας νομικά συστήματα, ακόμη και το, το, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρους το ISDS. Ευχαριστώ με τη σημερινή ακρόαση να ε, επισημάνω ότι υπήρξε και δημόσια διαβούλευση για το θέμα του ISDS και στη διαβούλευση αυτή συμμετείχαν ε, οι περισσότεροι πάρα πολλοί πολίτες. Ένα ιστορικό αποτέλεσμα για την δημοκρατία στην Ευρώπη. Όμως, επειδή δεν ήταν αρεστό το αποτέλεσμα, ε, προτιμήσατε να, και όπως ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους δεν τη η απόφαση να διαγραφεί το ISDS από τη συμφωνία TTIP. Τώρα μιλάμε για το πώς θα το βελτιώσουμε, θα το προσαρμόσουμε και θα το τροποποιήσουμε. Ήθελα να, ρωτη... ρωτήσω αν μετά από αυτές τις τροποποιήσεις θα ξαναζητήσουμε τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών για αυτό το μηχανισμό, το ISDS που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην ε, συνθήκη. Για να, λύσουμε, για να αναλύσουμε επί της ουσίας το όλο θέμα, το μόνο δεδομένο που σήμερα διαθέτουμε, τη συμφωνία με τον Καναδά, πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή δεν ευλήθηκαν σε καμία ε, περίπτωση οι αμφιβολίε για τους διαιτητέ, ούτε επί τη ουσία οι υποθέσεις. Οι δικηγόροι θα έπρεπε να ε, αναστέλουν προσωρινά τι δικηγορικές του δραστηριότητε. Έπειτα οι διαιτητέ, σε περίπτωση διαφωνία μεταξύ των μερών, τι θα κάνουν. Ένας ανώτατο υπάλληλο, ένα ανώτατο τέλεχος του, Παγκόσμια Τράπεζα ουσιαστικά καθορίζει το τι θα γίνει. Ε, με, ένας, με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι πολύ κοντά στα αμερικανικά συμφέροντα. Πώ θα έχουμε λοιπόν τη βεβαιότητα ότι υπάρχει ανεξαρτησία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν τα έκανε. Θέλει να μα κάνει να πιστέψουμε ότι τα εθνικά δικαστικά συστήματα δεν εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών επενδυτών. Πιστέψτε με, κυρία Επιτροπέ, εγώ έρχομαι από μια χώρα που δεν μπορεί να κρύψει κάποιε ελλείψει ε, και παραθυράκια στο δικαστικό του σύστημα. Ακόμη όμω και αν τα εθνικά μα δικαστήρια δεν είναι τέλεια, ε, ούτε τα συστήματά μας το ίδιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ε, αρκεστούμε σε ένα σύστημα που είναι ακόμη πιο ελαττωματικό. Θα πρέπει οι εσωτερικές προσφυγές να παραδεχτείτε ότι εφόσον πλέον δεν γίνονται θα είναι στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Τα εθνικά κράτη άλλωστε δεν έχουν ε, το ίδιο δικαίωμα πρόσβαση στο ίστιες. Λέτε ότι το δικαίωμα του ρυθμίζει θα εξασφαλίζεται, αλλά μόνο στο προήμιο και όχι στο κεφάλαιο για τις επενδύσεις και ολοκληρώνω πολύ σύντομα. Ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί διαμορφωθεί η πρότασή σας δεν λέει ε, ε, ότι δεν μπορούν οι διαιτητές να αποφασίσουν πρόστιμα δισεκατομμυρίων εις βάρος κάποιου κράτους. Ε, άλλωστε αυτό δεν ε, θα αποτελέσει, μόνο το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει φραγμός για την νομοθετική δραστηριότητα. Είναι σκάνδαλο κυρία Επίτροπε, είναι σκάνδαλο το SDS, αλλά σας συγχαίρω γιατί ένα σκάνδαλο καταφέρετε να το πιάσετε και να το κάνετε κουβέντα. Συγχαρητήρια για αυτό το κατόρθωμα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλές από τις ε, προτάσεις που αναφέρετε κυρία Μάλμστρο είναι πάρα πολύ θετικές και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο πατρίστες ήθελα να κάνω γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί όλες οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του ISDS κινούνται προς την δημιουργία ενός μόνιμου δικαστηρίου. Γιατί αυτό το παραπέμπεται σε μια διεθνή συμφωνία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ, γιατί η Δάλος θα ήταν απίθανο και θα μας καθυστερούσε πολλά χρόνια. Γιατί δηλαδή να μην κάνουμε το ίδιο για τη ΣΥΠΑ και να ισχύει φυσικά αρχικά μόνο για τη ΣΥΠΑ και μετά να κοιτάξουμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Για το ΣΕΤΑ τώρα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να λέμε ότι θα αλλάξει αυτό και λίγο η Συμφωνία ΣΕΤΑ. Είναι θέμα αξιοπιστίας, ελλείμματος αξιοπιστίας, το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Γιατί δεν ε, έχουμε και χρονικά τη λογική και ξέρουμε ότι πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις ε, έχουν έδρα στον Καναδά και έτσι μπορούν να γλιτώσουν από διάφορα στοιχεία τέτοια. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Δεν αποκλείεται αυτό αν υπάρχουν σχετικές εμπορικές δραστηριότητε. Γιατί λοιπόν δεν αντιμετωπίζετε επιθετικά το θέμα αυτό και δεν λέτε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα προς την κατεύθυνση που αναφέρετε γιατί το ρίσκο και οι συνέπειες του ρίσκου που συνεπάγεται το άνοιγμα του πακέτου είναι πολύ μικρότερο από το να αποτύχει συνολικά το ISDS. Και νομίζω ότι και η πολιτική ευθύνη βαρύνει ιδιαίτερα την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Σχέλνερ. Ευχαριστώ. Αν δεν έχει σπάσει, μην το διορθώνετε. Παρακολουθώ το θέμα εδώ και πολύ καιρό. Και πραγματικά δεν βλέπω τα προβλήματα προσπαθώ να παρουσιάσω Από τη δεκαετία του 50 είχαμε 600 περιπτώσεις. 31% τι έχασε το κράτος. Και ουσιαστικά ήταν καταγγελίες ε, συμβολέων και αδειών και ήταν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως ευρωπαϊκές ε, που ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι και εμείς έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ε, διμερών επενδυτικών ε, συμφωνιών στον κόσμο και δεν έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών και άλλων προδιαγραφών. Αν δεν έχει σπάσει λοιπόν, μην το προσπαθείτε να το διορθώσετε. Επίσης, τι γίνεται με την αρχή ο χαμένος να πληρώνει για παράδειγμα για την καταβολή των δικαστικών δυτικών εξόδων. Και μάλιστα είναι σκαδαλώδες που ότι χθε εμποδίσαμε την ε, δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραμμίσει να υπογράψει την συμφωνία ISDS στην συμφωνία στην CITRAL, δηλαδή στην Επιτροπή του Ενωμένου ΕΕ για το Εμπορικό Δίκαιο. Επίσης, τι γίνεται με το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Νομίζω από τη στιγμή που έχουμε χάσει μόνο 31% των υποθέσεων, είναι προς το συμφέρον μας να έχουμε μια τέτοια δυνατότητα. Και επαναλαμβάνω, κυρίως οι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν. Επίσης θα πρέπει να αποτρέπουμε τους νομοθέτες από το να κάνουν το έργο τους. Γιατί πρόκειται για νομοθεσίες που απαλωτριώνουν χωρίς αποζημίωση, που κάνουν διακρίσεις, δεν θα αποδυναμώσουμε το σύστημα με τη μεταρρυθμίση αυτή. Θέλουμε ένα εύρυθμο νομικό σύστημα, ισχυρό και αυτή τη μάχη θα πρέπει να δώσουμε παντού. Δεν μπορούμε να λέμε ότι απλώς έχουμε εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος θα πήγαινε, θα εμπιστευόταν ένα δικαστήριο στο Τενεσί. Ούτε εσείς φαντάζομαι. Επίσης, έχουμε χώρες ε, σε θέσεις 130 ε, και 136 στην παγκόσμια κατάταξη δικαστικών συστημάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η κυρία Σκακέλε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε κύριε Επίτροπε, μας παρουσιάσατε τα σχέδιά σας, τις προτάσεις σας, που θα έλεγα ότι σίγουρα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ε, χτυπάν το κακό στηρίζεται, δεν φτάνουν στον πυρήνα του προβλήματος. Δεν είχαμε ουδέποτε ε, μια εις συζήτηση για το αν θέλουμε πραγματικά το ISDS. Η συζήτηση ήταν τι είδους ISDS θέλουμε και η διαβούλευση ήταν επί των μεταρρυθμίσεων που προτείνεται στο ISDS. Το θέμα είναι να έχουμε συζήτηση επί της αρχής. Θέλουμε καταρχήν ISDS ή όχι. Τώρα για πρώτη φορά έχουμε τέτοιες αρμοδιότητες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα ή όχι. Γιατί τώρα θα αποφασίσουμε θα να το φορτωθούμε μέχρι ε, την Δευτέρα παρουσία ή να απαλλαχθούμε από αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη και βασική ε, ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας. Αν θέλουμε πραγματικά ένα τέτοιο σύστημα. Είδαμε τις ε, προτάσεις σας για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά άλλο είναι το βασικό ερώτημα. Αν Κατά βάση χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και εντό και εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δημόσια ευρωπαϊκή συζήτηση. Αναφέρθηκε και το Διεθνέ Δικαστήριο. Μπορούμε να το συζητήσουμε, ίσως θα ήταν ενδιαφέρουσα πρόταση. Η κόκκινη γραμμή είναι να συμπεριλαμβάνονται και αγωγέ κατά των επενδυτών, γιατί πολλέ καταχρήσει ε, διαπράττονται από του ίδιου του επενδυτέ. Οπότε θα πρέπει να περιλάβουμε σε τέτοιε διατάξει και τι υποχρεώσει των ίδιων των επενδυτών. Τώρα το να πούμε στο DTIP ότι αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να επιδιώξουμε την, ζήτηση, την δημιουργία ενός μόνιμου διεκτικού δικαστηρίου και εντωμεταξύ λέμε όχι στο SDS. Γιατί να μην προτείνουμε και κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τη ΣΥΤΑ, τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά, είπατε ότι διεκπαιρεώθηκε, ότι δεν έχουμε περιθώρια επιλογών. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν κάποια πράγματα ή όχι. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, διατήρηση του δικαιώματος του νομοθετή, ναι, του ρυθμίζει για τις ε, κυβερνήσεις, τι ακριβώς διατύπωση θα χρησιμοποιήσετε στο άρθρο. Κύριος Κάσπαρη. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι κατέστη εκ νέου σαφές ότι αν ε, δεν θέλουμε να ισχύει το δίκαιο του πιο ισχυρού, αλλά το δίκαιο του δικαίου, θα πρέπει να ρυθμίσουμε την παγκοσμιοποίηση. Διάφορα έχουμε σχολιάσει. Οι διεθνεί συμβάσει δεν είναι εφαρμόσιμε από τα εθνικά δικαστήρια. αφού το γράφουμε σε κάθε συμφωνία ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι βασικό ζήτημα. Και καλώς γίνεται έτσι. Σχετικά με τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από συμφωνίες με τρίτα κράτη, καλύτερα είναι να διευκρινίζονται αυτά με τρίτα δικαστηρία. Παρά το γεγονός, παρά την περίπτωση να έπρεπε να, να προσφύγουμε σε ένα κομμουνιστικό δικαστήρια μιας κομμουνιστικής χώρας. Αν σκεφτούμε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια που είχαμε την προσφυγή ε, του αεροστόλου και η Airbus, η Airbus ε, είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει διάφορες, διάφορα κόλπα. Αν λοιπόν αυτό δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση δαπών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ. Κάτι άλλο. Ακούσαμε ότι η συμφωνία με τον Καναδά είναι παλιά η συμφωνία, αυτή η εμπορική συμφωνία. Δεν ισχύουν όμως ε, τα όσα ισχύουν στο παρελθόν με τον Καναδά σε σχέση με τις 1.400 άλλες αντιμερείς ε, Διεθνής Συμφωνίας. Η συμφωνία με τον Καναδά αποτελεί ένα τεράστιο βήμα βελτίωσης. Γι' αυτό λοιπόν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με τη συμφωνία με τον Καναδά ε, πραγματικά φυσικάζονται πολλές από τις ανησυχίες που είχαμε από άλλες διεθνείς συμφωνίες. Κάτι άλλο. Θέλουμε να έχουμε πολιτικό περιθώριο ελιγμού. Και είναι καλό που το αναφέρουμε αυτό και πάλι σήμερα, αλλά θα ήθελα να κάνω κριτική σε δύο σημεία και να κάνω και προτάσεις. Το πρώτο το θέμα της δυνατότητας αναθεώρησης. Και εγώ θα επιθυμούσα να υπάρχει. Αλλά να σκεφτούμε εάν σε τελική ανάλυση αυτό θα είχε ωφέλη για μας ως νομοθέτες. Γιατί ω τώρα μόνο 25% των περιπτώσεων δικαίωσαν τους επενδυτές. Άρα ουσιαστικά δίνουμε άλλη μια δυνατότητα αν ε, καταδικάζεται ένα κράτος γιατί να μην ζητήσει αναθεώρηση. Να σκεφτούμε. Και κατά τρίτον για τα δικαστήρια. Και εδώ, αν δημιουργηθούν διεθνή δικαστήρια, μπορώ να φανταστώ αυτό στο μέλλον να γίνει. Δεν θέλω όμως να γίνει κάτι τέτοιο υπερβολικά γρήγορα και να μην εισαχθεί αυτό κατευθείαν στην Αμερική. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Αμερική, θα πρέπει να το συζητήσουμε και με άλλου να υπάρχουν όσο πιο, πολύ, όσο πιο πολλέ χώρε γίνεται. Και προφανώ εγώ προτιμώ κάποιου ε, ιδιωτικού δικαστέ, ιδιωτικού δικαίου, παρά κάποιου που θα του έχουν διορίσει δικτατορικά καθεστώτα η κομμουνιστικά καθεστώτα. Η κυρία Ρέντιν και μετά η κυρία Αρένα. Well, thank you. Ευχαριστώ. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα την Επίτροπο Μάλμστρομ. Γιατί αυτά που μας είπε σήμερα είναι πολύ σημαντικά και κάνει ένα πολύ σημαντικό άνοιγμα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί είπε ότι χρειαζόμαστε βραχυπρόθεσμα, άνοιγμα και μεταρρύθμιση και μέσω πρόθεσμα ίσως και πιο ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση. Για παράδειγμα, εγώ είχα προτείνει τη σύσταση ενός μόνιμου ε, διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Βέβαια, η σύσταση ενός διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου δεν είναι βραχυπρόθεσμη λύση, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά σε τελική ανάλυση αυτό θέλουμε. Όχι φυσικά κομμουνιστικού τύπου διεθνέ δικαστήριο, αλλά ένα διεθνέ διαιτητικό δικαστήριο που θα διέπεται από το κράτο δικαίου. Και σίγουρα αυτό που είναι κατάλληλο είναι ο παλιός μηχανισμός με τις 1.300 διαφορετικές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Σίγουρα η συμφωνία με τον Καναδά συνιστά ένα άλμα πρόοδο και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε διαπραγματεύσεις για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία. Γιατί από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει, θα πρέπει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Πάκτα σουν σερβάντο. Δεν θα πρέπει να αναλάβετε στην πρωτοβουλία και να ξαναρχίσετε διαπραγματεύσει. Αλλά να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που έχουμε και με έναν εταίρο που είναι πολύ οικείος να φροντίσουμε να προτείνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μερικές ήδη έχουν προταθεί ως τροφή για σκέψη, να τις αναλύσουμε διεξοδικά και ίσως αυτή θα ήταν και η απάντηση στις α, α, χιλιάδες ερωτήσεις που μας έκαναν οι πολίτες, γιατί πραγματικά ξεκίνησε η διαδικασία ε, και έγινε μια διαφανής διαβούλευση για το θέμα αυτό. Και γιατί να μην ε, έχουμε και ένα δευτεροβάθμιο σώμα που θα ήταν ίσως το πρώτο βήμα για ένα διεθνές διεθνικό δικαστήριο. Και θα μπορούσαμε να είναι ήδη μια ε, τέτοια ε, αρχή, μεσοπρόθε, με, μια μάλλον προσωρινή λύση που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο DTIP είναι το Διεθνές ε, Δικαστήριο που ήδη υπάρχει οικονομικά θέματα των Ηνωμένων Κυρία Αρένα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, προσπιζόμενοι Μάλλον αυτο η αρχή που, που είναι ότι όλοι οι επενδυτές ασχέτως της εθνικότητά τους θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και ένα σύστημα δικαστικό αμερόληπτο, δίκαιο και ε, ανεξάρτητο. Είναι αμερόληπτο και δίκαιο το ευρωπαϊκό σύστημα. Το αμερικανικό είναι έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι ισχύει. Όμως έπειτα το θέμα είναι τι θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα σύστημα προστασίας των επενδυτών. Πρώτα απ' όλα να ευνοήσουμε τις επενδύσεις των ε, ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν τέτοιε επενδύσεις. Ο κύριος Πρόεδρος είπε το πρωί ότι η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα που έχει αποφεληθεί από αυτές τις επενδύσεις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και ότι δεν υπάρχει ISDS. E ISDS. Δεν υπάρχει τους μηχανισμό. Δεν σημαίνει ότι αυτό κινείται τι επενδύσει. Έπειτα θέλουμε να προστατεύσουμε του επενδυτέ που πάνε στι ε, ΗΠΑ τους δικούς μας. Η ε, απάντηση είναι ότι ε, έχουμε επενδυτές στις ΗΠΑ σε ό, από όλα τα κράτη και είναι προστευμένοι. Τρίτον, θέλουμε να προσπαθούμε το δικαίωμα το ρυθμίζει. Αυτό, με συγχωρείτε, το μηχανισμός ISDS δεν το, δεν το επιτυγχάνει. Με αυτό λοιπόν, ε, με αυτή την κατάσταση που ισχύει σήμερα και το επιχείρημα, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ISDS στο πλαίσιο του TTIP. Διότι ακριβώς το ISDS δεν δυσφαλίζει το δικαίωμα το ρυθμίζει και μάλιστα θα το αποδυναμώσει, θα το υποβαθμίσει. Επίτα μας λέτε το επιχείρημα ε, ότι εννέα χώρες, ε, νέα κάτι μέλη έχουν SDS ε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επειδή εννέα κάτι μέλη έχουν SDS πρέπει να ευθυγραμμιστούν 28 με τους υπόλοιπους 9. Ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Δεν συμφωνώ. Τρίτον, Α δεχτούμε ότι έχουμε δικαιοδοσίε που κάποιε φορέ δεν λειτουργούν τέλεια, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αλλά όταν βλέπουμε το κόστο του ISDS για μία μικρομεσαία επιχείρηση, θα είναι απαγορευτική πρόσβαση για το κόστο. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό το επιχείρημα, δεν ευσταθεί. Συμφωνώ μαζί σα όμω σε κάτι άλλο, κυρία Μάλστρομ, ότι πρέπει να επεξεργαστούμε ένα μηχανισμό ISDS για το μέλλον, όχι για το TTIP. Για το μέλλον, ναι. Ένα σύστημα που να είναι πολύ πιο δίκαιο, πολύ πιο ισόρροπο και βρίσκω ότι οι προτάσει που κάνετε σήμερα είναι προτάσει που είναι ενδιαφέρουσε, θα μπορούσαμε να τι επεξεργαστούμε αλλά πρέπει να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή. Όχι μόνο για τη συμφωνία TTIP, αλλά γιατί εμ, ε, επιμένοντας το ISDS θα δικηβεύσουμε ολόκληρο το TTIP. Ας ε, επεξεργαστούμε καλύτερα με το πώς θα επιλύονται οι διαφορές εκτός του TTIP και είμαστε έτοιμοι και στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε όσο θέλετε αυτό. Ευχαριστούμε. Μορέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, γιατί το μηχανισμό ISDS προκαλεί τόση συζήτηση. Και γιατί υπήρξαν τόσε αρνητικέ απαντήσει στο σα. σας. Ε, ενώ προσπαθήσατε καταρχά να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο αυτών των αρνητικών απαντήσεων. Τώρα ήρθατε ενώπιον με προτάσεις, καλό είναι και αυτό, γιατί καταλάβατε ότι και εμεί ε, και εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με, το, με την κατοική διάσταση του θέματος ως το ESDS. Δεν είναι το μόνο πρόβλημά μας με τη συμφωνία TTIP, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μας ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι προσπαθούμε να δώσουμε το πάνω χέρι στους επενδυτές και ξεχνάμε τους πολίτες ή το κράτη. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια καχυποψία σε σχέση με την ιδιωτική δικαιοσύνη. Ε, υπόθηκε επανειλημμένος. Και ιδίω το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που ε, θα υπάρχει εφόσον οι ιδιώτες ε, εμπλέκονται στο θέμα αυτό. Και βεβαίω είναι το θέμα πώ θα ορίσουμε και τη σύγκρουση συμφερόντων. Όταν σα ακούμε, όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι τρόπον τεινά το SDS είναι απερχιωμένο και πεπαλαιωμένο. Όμω, αντί να ασχοληθούμε με τι σημερινέ προτάσει πρώτα απ' όλα, α απαντήσουμε πρώτα στην ερώτηση. Το χρειαζόμαστε απαραίτητο στο πλαίσιο τη Ιθλανδική συνθήκη. Είναι απολύτω απαραίτητο. Ποιο το ζητά. Διότι εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσο σχετισμό στατιστικό ε, με την, για την παρουσία του ISDS και την αύξηση των επενδύσεων από τη μια ή την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι κάτι στο οποίο δεν έχουμε επιμείνει ακόμα αρκετά είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, αποτρέπονται από το να λάβουν δημόσια μέτρα ε, από φόβο μήπως προσφύγουν αντίον τους οι επιχειρήσεις. Ε, εκτός είναι κάτι καλά, αν δεν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπατε. Και τρίτη ε, παρατηρήση για τη ΣΕΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά. Λέτε εδώ ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί, έχει περατωθεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, και ταυτόχρονα ε, λέτε ότι από αύριο θα φτιάξουμε ένα φανταστικό SDS, τελείω αναθεωρημένο. Μα κοιτάξτε, εάν δεχτούμε την συμφωνία ΣΕΤΑ ως έχει, με το μηχανισμό SDS που δεν λειτουργεί καλά. Αύριο γιατί οι Αμερικανοί να μην έρθουν να μα πούνε ότι με τον Καναδά έχετε κάτι που δεν λειτουργεί και τόσο πολύ καλά ή λειτουργεί έτσι και έτσι. Εμά γιατί μα επιβάλλεται μια μεταρρύθμιση του συστήματο. Ε, η συμφωνία ΣΕΤΑ ε, θεωρήθηκε μια καλή συμφωνία. Εφόσον εγκρίθηκε όμω, σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε θετική απάντηση και στο TTIP, ενώ είναι πάρα πολύ τα ερωτήματα που παραμένουν εκκρεμή. κυρία Σαρασνόβα και μετά ο Σίλβα τελευταία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε και μας παρουσιάσατε τις τελευταίες σας προτάσεις για το μηχανισμό ASDS. Μιλήσατε γενικά για διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ χωρών, αλλά η Τσεχία, η πατρίδα μου, έχει περίπου 80 επενδυτικές, διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και μάλιστα έχουμε τέτοια διμερή επενδυτική συμφωνία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι κάπως απερχιωμένη και θέλουμε να την εξυγχρονίσουμε. Και πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος εξυγχρονισμού τέτοιων συμφωνιών είναι με μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση και έναν ενιαίο μηχανισμό ASDS. Όχι μόνο για την TTIP, αλλά και για τις μελλοντικέ μας εμπορικές συμφωνίες. Και για την TTIP έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε μια τέτοια συμφωνία και ένα μηχανισμό ISDS για τις εταιρείε μας. Γιατί όπως είπατε, οι διεθνείς συμφωνίες δεν εφαρμόζονται από τα ε, αμερικανικά δικαστήρια. Και αυτό είναι μειονέκτημα για μας. Και Τώρα, η ιδέα για ένα μόνιμο διευθυντικό δικαστήριο είναι εύστοχη, αλλά όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ε, προϋποθέτει μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν πρόκειται να γίνει εν μία νυχτή. Εμείς όμως ήδη από τώρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε τις διατάξεις ISDS και να τις συμπεριλάβουμε στην DTIP. Συμφωνώ με την πρότασή σας που ακολουθεί τη σωστή πορεία και πολύ ευχαρίστω θα συμμετέχω και στη συνέχεια στη συζήτηση. Ο κύριος Σίλβα, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σας και για την συζήτηση που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε. Έχω μία ερώτηση, μία διευκρίνηση θα ήθελα. Πόσο φιλόδοξη θα είστε και πόσο θα βελτιώσετε τις διατάξεις ISDS στη ΣΥΤΑ. Γιατί παρά τις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που έγινε για τη ΣΥΤΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς αυτό δεν ήταν αρκετά καλό και γι' αυτό χρειάζονταν ε, αλλαγές και βελτιώσεις. Οπότε έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα εδώ. Δεν βλέπω πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα μπορέσει να εγκρίνει μία εμπορική συμφωνία όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν είναι αρκετά καλή αυτή η εμπορική συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσετε με τους Καναδούς εταίρους μας ε, εναλλακτικέ λύσεις. Να γίνουν κάποιες ε, βελτιώσεις ε, στο ISDS. Είπατε ότι γίνεται αυτό και είπατε προτάθηκε και ένας δευτεροβάθμιος μηχανισμός διατησίας ή η ρήτρα απανεξέτασης για το μέλλον. Θέλω όμως διευκρινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα σε ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να συνεχίσει τις ε, διαπραγματεύσεις με τους Καναδούς και πόσο μακριά μπορεί να πάει. Ιδιαίτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Γιατί μόνο είναι θετική αυτή η απάντηση σε ερωτήσει. Μιλούμε για ένα πραγματικό άνοιγμα και έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο κεφάλαιο αυτό. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Επίτροπο για να απαντήσει. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει και για τα σχόλια. Μάλιστα μερικά επικαλύπτονται, γι' αυτό και προσπάθησα να τα ομαδοποιήσω για να εξοικονομήσω και λίγο χρόνο. Πολλοί ε, είστε της γνώμης ότι το ISDS ε, είτε με την παρούσα του μορφή είτε με περαιτέρω αλλαγές ε, είναι περιττό. Υπάρχει όμως ήδη αυτό. Έχουμε νέα τέτοιες ε, συμφωνίες ε, με τις ΗΠΑ Πολιτείες, ε, και με την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερο στον κόσμο. Δεν μπορούμε να τις διαγράψουμε μία μονοκοντιλιά αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχουν ήδη. Και είναι τμήμα της εντολής που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα αποτελεί και προτεραιότητα των Ηνωμένων ρήτρα ISDS θα περιληφθεί σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες. Στην ε, Διευρυνική συμφωνία επίσης υπάρχουν τέτοιες ρήτρες ISDS. Οπότε, αν ε, ε, καταργήσουμε εμείς μια τέτοια ρήτρα, θα βρεθούμε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τον Καναδά, η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη ρήτρα στην συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αλήθεια είναι ότι οι διεθνείς συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο ε, με βάση την Αμερικανική νομοθεσία δεν ε, θεωρούνται ως δίκαιο εφαρμοστέο. Ο κύριος Φιέλερ μας έδωσε στατιστικές στοιχείες που είναι γνωστές και είδατε τις περισσότερες περιπτώσεις τις χρησιμοποίησαν ευρωπαϊκές εταιρείες αυτές τις ε, διεξόδους και μάλιστα μικρομεσαίες για να ε, διαφυσβητηθούν διακρίσεις, ε, ξαφνικές αλλαγές αδειών, δημέψεις, κατασχέσεις. Ε, είναι σημαντικά ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν χιλιάδες ή εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτές τις εταιρείε από τα σπάνια αυτά φαινόμενα που υπάρχουν όμως. Όντως είναι σπάνιες περιπτώσεις και για αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις θέλουμε να προστατεύσουμε τις εταιρείε μας για να ελαχιστοποιήσουμε την καταχρηστική εφαρμογή του συστήματος και γι' αυτό έχουμε και μια συσταλτική περιγραφή. Και πολλά από αυτά τα θέματα καλύφθηκαν και από τη ΣΕΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά. Αν διαβάσετε τη συμφωνία αυτή, διαπιστώνετε ότι ήδη υπήρχαν πολλέ μεταρρυθμίσει. Την αρχή ο, αυτός που έχασε πληρώνει. Αυτό υπάρχει ήδη στο ΣΕΤΑ. Φυσικά, αυτό που έχασε την δίκη καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Ισχύει αυτό και στη ΣΕΤΑ και έχει και ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα διεθνή δικαστή, διεθνές δικαστήριο, μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο. Καλή ιδέα, αλλά ήμουν ειλικρινή από την αρχή και είστε και εσείς ρεαλιστές. Δεν πρόκειται να γίνει εν μία νυχτή, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Και πρέπει φυσικά να βρούμε συμμάχους και πώς θα λειτουργήσει ένα τέτοιο δικαστήριο, πώς θα χρηματοδοτηθεί, ποια θα είναι τα μέλη, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το μόνιμο δικαστήριο και να αναβάλουμε το επίγον ζήτημα που είναι το TTIP και το ISDS. Γιατί περιμένουμε και άλλες χώρες, η Ιαπωνία στη σειρά και άλλες. Θα πρέπει να βρούμε λύση λοιπόν σε αυτό το θέμα, φυσικά κάνοντας ένα άνοιγμα για το μέλλον. Και οι υπηρεσίες μου, σας είπα, ήδη διερευνούν την δυνατότητες ε, σύστασης ενός διεθνούς μηχανισμού. Τώρα, Φυσικά υπάρχει το Διεθνέ Κέντρο Επίλυση Διαφορών Επενδυτών τη Παγκόσμια Τράπεζα και υπάρχει και όλε οι χώρε δεσμεύονται. Τώρα, δευτεροβάθμια διατησία. Είτε θα είναι ένα μόνιμο ε, σώμα με βάση, υπό την αίγυδα του ΠΟΕ και θα έχουμε, ήδη έχουμε πάνελ στα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν μια πιθανή λύση. Και επίσης ε, θα είχε νόημα σε ένα ε, εύρωστο ένομο σύστημα με αμοιβαιότητα και νομιμοποίηση να υπάρχει ένας μηχανισμός δευτεροβάθμιας, όχι μόνο για τις εταιρείε, αλλά και για τα κράτη-μέλη, να υπάρχει δυνατότητα ε, έφεσης. Πολλοί ρωτήσατε για τη ΣΕΤΑ. Η ΣΕΤΑ είναι μια συμφωνία που έχει ολοκληρωθεί. Ανα... Μάλιστα στις 27, 26-27 Νοεμβρίου αναγγέλθηκε ε, και από τον ε, Καναδό Πρωθυπουργό και από τις 28 χώρες μέλη. Κάποιες ε, νομικές ε, τελειοποίησεις θα γίνουν και μετά θα περάσει στη μετάφραση συμφωνία. Φυσικά θα συζητήσουμε με τους Καναδούς και τους Αμερικανούς εταίρους, αλλά Φυσικά, πρώτα θα πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας και να συνεννοηθούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βρούμε εμείς μια λύση. Και αν η πλειοψηφία τουλάχιστον συμφωνήσει για το πώς θα προχωρήσουμε, τότε θα το συζητήσουμε και με τους Αμερικανούς και με τους Κανάδους φίλους σε πλήρη διαφάνεια ώστε να γνωρίζετε τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να ξεκινήσω τις διαπραγματεύσεις με τους Καναδούς πριν α, ε, ε, μάθω τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε αν στο μελλοντικό ISDS υπάρχουν κάποια θέματα που στη φάση της νομικής ε, τελειοποίησης θα μπορούσαν να περάσουν και στην Καναδική Συμφωνία. Αλλά χωρίς να ξαναρχίσουμε διαπραγματεύσεις ε, ε, της συμφωνίας με τον Καναδά. Καμία χώρα επίσημα δήλωσε κάτι τέτοιο. Γιατί έστω και ένα κεφάλαιο να ανοίξουμε, να είστε βέβαιοι ότι οι Καναδοί θα ανοίξουν δεύτερο κεφάλαιο και μετά δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Κάτι που θα είναι κακό και για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για την αξιοπιστία μας ό,τι αφορά τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τη σωστή ισορροπία και όχι άνοιγμα νέων διαπραγματεύσεων. Χρονοδιάγραμμα. Το ζήτησαν αρκετοί. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη συζήτηση. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχιστεί και σε κυβερνητικού σχηματισμού. Με τα χαράς λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα και να συζητούμε. Το Συμβούλιο Εμπορίου την ερχόμενη εβδομάδα, τα άτυπα συμβούλια δικαιοσύνη θα τα συζητήσουν, θα τα δούμε και εσωτερικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην Άνοιξη. Δεν έχω συγκεκριμένε ημερομηνίε δυστυχώ. Αλλά καλά θα ήταν να το ολοκληρώσουμε το θέμα, διότι όπω είπατε υπάρχουν και άλλα πολύ ε, καυτά ζητήματα, πιεστικά ε, για το τι που πρέπει να συζητηθούν. Μέσα στην Άνοιξη λοιπόν ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόταση και πρέπει να συζητήσουμε ακριβώ το πότε. για τη Γιούν την Επιτροπή Ηνωμένων Πολιτειών για το Εμπορικό Δίκαιο, Έχετε δίκιο κύριε Χέλνερ, πρέπει να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη διαφάνεια. Για το δικαίωμα του ρυθμίζει ε, η πρόταση στην ε, Καναδική Συμφωνία αναφέρεται στο προήμιο όντω. Η πρόταση είναι να περάσει πλέον στο σώμα του κειμένου, του νομικού κειμένου. Και Νομίζω ότι ρητό διαφυλάσσεται το δικαίωμα του ρυθμίζει στο ίδιο το σώμα του κειμένου, έτσι όπω προτείνεται. Πρόεδρε, νομίζω ότι λίγο πολύ κατάφερα να καλύψω τις ερωτήσεις, γιατί τις ομαδοποίησα ανά θέμα. Να με συγχωρείτε αν κάτι μου διέφυγε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Σίγουρα θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε και απαντήσατε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ολοκληρώνουμε έτσι το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Να αρχίσω ευθύ αμέσω με το σημείο 7. Σημείο 7 λοιπόν, TTIP. Ποια τα ωφέλη για τους Ευρωπαίους. Ίσως να μας δίνατε 2-3 λεπτά, λέει η Επιτροπός. Εάν υπάρχουν μετακινήσεις, να είστε γοργοί και ήρεμοι. Hat es den entsprechenden Austausch... Μάλιστα, αν ολοκληρώθηκαν τα σχετικά τριγαδάκια. Da möchte ich aber wirklich jedem bitten, ruhig zu sein. Please. Σας παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία για να προχωρήσουμε. So, Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόασή μας. Έχουμε διοργανώσει μια σειρά ακροάσεων για διάφορα τμήματα της ε, διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία TTIP. Συμφωνήσαμε, συζητήσαμε καταρχάς το θέμα του ISDS και σήμερα θέλουμε να εστιαστούμε στο συγκεκριμένο θέμα του τι Οφέλη έχει για τους Ευρωπαίους η συμφωνία TTIP. Θα φαντάζεστε άλλωστε ότι σχεδόν ε, καθημερινά έχω διάφορες ε, εκδηλώσεις για το TTIP και αυτή η ερώτηση εγκυμένα ακούγεται κάθε μέρα. Κάποιος πολίτης παίρνει το λόγο και λέει πείτε μου τι ωφέλη έχει για μένα συγκεκριμένα η συμφωνία TTIP. Αυτό λοιπόν αποτελεί το θέμα της σημερινής ακρόασης σε προσωπικό επίπεδο ή και σε ομαδικό επίπεδο ιδιωτών. Τι ωφέλη συνεπάγεται η συμφωνία TTIP και χαίρομαι ιδιαίτερος που η Σεσίλια Μάλμστροπ η αρμόδια επιτροπή για θέματα εμπορίου θα μας κάνει μια εισαγωγή στην ε, ακρόαση αυτή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Να περάσουμε από το μηχανισμό ESDS στην ε, γενικότερη εικόνα. Σα ευχαριστώ που οργανώσατε αυτό το, αυτή την εκδήλωση. Είναι τεράστια σημασία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον πολιτικό κόσμο, αλλά και μεταξύ των πολιτών, των ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη και προσπαθώ, θα προσπαθήσω να πω όσο πιο πολλά μπορώ. Ε, είναι τεράστιο ενδιαφέροντος. Ε, είναι πολλά τα ερωτήματα και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το πάνελ που έχετε προβλέψει σήμερα το απόγευμα. Απλώς μια σύντομη εισαγωγή εδώ. πολιτική, τακτική μου ήταν όταν ανέλαβα αυτή τη θέση εδώ και 4,5 μήνες ότι η εμπορική πολιτική να ε, προσανατολίζεται προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια για το διάλογο ώστε οι άνθρωποι να συμμετέχουν και να ε, έχουν ε, πλήρη ανάληψη ευθύνη και να εκφράζουν τις απόψεις τους και βεβαίως και για τις εταιρείες οι εταιρείε, οι επιχειρήσει, είναι αυτέ που διαμορφώνουν το περιβάλλον, ε, όπου προσπαθούμε να άρουμε για αυτέ του φραγμού για τι εξαγωγέ του. Και βεβαίω επηρεάζουν τον πραγματικό κόσμο. Οι εταιρείε γνωρίζουν ποιοι είναι οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν και τι είδου οικονομική δυνατότητα μπορεί να ε, προσφέρει το εμπόριο. Σε μια δεύτερη φάση βεβαίω θέλουμε περισσότερε θέσει εργασία και περισσότερο ωφέλη και περισσότερο κέρδο και οικονομικό κέρδο για του πολίτε. Και βεβαίω ε, υπάρχουν άτομα με πολλέ διαφορετικέ ιδιότητε, ενώσει καταναλωτών, συνδικαλιστέ οργανώσει, περιβαλλοντικέ οργανώσει, ακτιβιστέ. Όλοι αυτοί είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων και η εμπειρία του είναι πολύτιμη. Μπορούν να μα μιλήσουν για τον ευρύτερο αντίκτυπο τη άρση των φραγμών στον τομέα του εμπορίου. Προσπάθησα να ακούσω όλε αυτέ τι απόψει και θέλαμε να δημιουργήσουμε μια σειρά από προτεραιότητες για την προστασία των καταναλωτών ώστε να διαφυλάξουμε ή και να ενισχύσουμε την νομοθεσία μας που την ε, εγγυάται. Έτσι έχουμε συνάψει τώρα τι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο θα κάνουμε και στο TTIP. Οι μέρημνε που άκουσα τώρα να εκφράζονται και οι ανησυχίε έχουν να κάνουν με το ότι οι διαπραγματεύσει δεν είναι αρκετά διαφανεί. Πολλοί αισθάνονται ότι για το TTIP υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες ε, και καλό θα ήταν να είμαστε τελείως ανοιχτοί. Ε, κανονισμός για τη διαφάνεια ε, ισχύει εντός της Ευρώπης, οπότε προφανώς πρέπει να ισχύει και διεθνώς. Γι' αυτό αναλάβαμε πρωτοβουλίες για να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις για εσάς, τα μέλη του Κοινοβουλίου, τις εθνικές κυβερνήσεις και το κοινό. Αυτό αυτό το ανοιχτό πνεύμα βελτιώνει την ποιότητα του διαλόγου φυσικά. Ε, κάνει όλους να καταλάβουν το τι κάνουμε. Πολλά είναι τα έγγραφα που ε, βρίσκονται στο διαδίκτυο ε, και νομικά κείμενα και σημειώματα τοποθετήσεως, τοποθετήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα σωρό άλλες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω είναι καθοριστική σημασία σε αυτό ε, γιατί τα ωφέλη όλες της συμφωνίας αρχίζουν να φαίνονται. Ε, να αναφέρω τρία από αυτά. Προφανώς να ενισχυθεί η οικονομία μας, η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησή μας και η φωνή μας παγκοσμίω. Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Το TTIP θα ωφελήσει του Ευρωπαίου γιατί θα ακουστεί η χειρότερα φωνή μα εκτό των δικών μα των συνόρων στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι οι πολιτικέ μα εκτό γίνονται εδώ ένα και περισσότερο σημαντικέ. Η παγκόσμια οικονομία με τι επικοινωνίε, την τεχνολογία, τι διεθνεί συναλλαγέ γίνεται όλο και πιο ενοποιημένη από τι κυβερνήσει. Απαιτούνται διεθνεί κανόνε τόσο για τα πρότυπα ασφαλεία ω τι κεφαλικέ απαιτήσει για τι τράπεζε. Αυτή η ε, ε, συζήτηση για τη διεθνή συνεργασία θα αυξηθεί στο μέλλον. Και επειδή συμβαίνει αυτό, το σχετικό μέγεθο τη ευρωπαϊκή οικονομία ε, στον κόσμο μειώνεται. Το ίδιο ισχύει για τι ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι και δύο πλευρέ θα έχουν λιγότερη επιρροή και λιγότερο βαρύτητα στο διεθνέ προσκήνιο, εάν δεν συνεργαστούν. Γι' αυτό ε, το ότι θέλουμε το ίδιο για του διεθνεί κανόνε, με αυστηρού κανόνε για το περιβάλλον, για του καταναλωτέ, για την υγεία, την ασφάλεια και άλλα θέματα, αυτό μα φέρνει πολύ κοντά και το TTIP επιτρέπει τη συνάρτηση αυτή τη συλλογιστική. Δηλαδή ενισχύει την εταιρική σχέση που έχουμε με τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα σωστό ρυθμιστικό ρεαλιστικό πλαίσιο για τα θέματα που θέλουμε να στήσουμε επιρροή και στο μέλλον. Αυτό είναι όφελο για του Ευρωπαίου πολίτε. Η δεύτερη κατηγορία όφελων έχει να κάνει με τη κυβέρνησή μα και ε, έχει να κάνει με το εξή. Η ρυθμιστική συνεργασία θα είναι στον καρδιά, τον πυρήνα του TTIP. Και οι ρυθμιστέ όταν συνεργάζονται κάνουν καλύτερε ρυθμίσει. Ε, ανταλλάζουν δεδομένα, ε, πληροφορίε. Υπάρχουν ρυθμιστικέ προκλήσει από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα μέχρι την ανατεχνολογία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μετωπίση τη αβεβαιότητα. Εάν λοιπόν συγκεντρώσουμε ε, τι γνώσει μα, θα έχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση για να προστατεύσουμε του πολίτε μα και να έχουμε υψηλότερα τα πρότυπα. Και έπειτα, εφόσον συνεργάζονται οι ρυθμιστέ, επιβάλλουν καλύτερα και του κανόνε. Οι αρχέ έχουν έναν ε, περιορισμένο αριθμό επιθεωρητών για να βεβαιωθούν ότι οι κανόνε γίνονται σεβαστοί. Η συνεργασία και από τι δύο πλευρέ για τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά και ένα σωρό άλλα θέματα, θα βοηθήσουν τα πράγματα. Οι κυβερνήσει επίση θα μπορούν ευκολότερα να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίε χρησιμοποιώντα συνετότερα το χρήμα των φορολογημένων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό. Αλλά και οι δασμοί, η μείωση των δασμών ε, θα κάνουν τα προϊόντα φθηνότερα, τα φάρμακα, τα ενδύματα, τα έπιπλα. Αυτό θα είναι εξοικονόμηση του χρήματο των φορολογουμένων. Αλλά είναι σαφέ ότι δεν θα υποβαθμιστούν τα πρότυπα ούτε για τα τρόφιμα, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την υγεία, ούτε για την ασφάλεια, ούτε για την προστασία των καταναλωτών με τη συμφωνία TTIP. Όλα όσα γίνονται για το TTIP, για την υπάρχουσα ευρωπαϊκή και αμερικανική νομοθεσία, θα φέρει σε ψηλότερο επίπεδο τα πρότυπα. Τίποτα από αυτά που θα κάνουμε δεν θα επηρεάσει το επίπεδο των προτύπων μας και οι επενδύσεις δεν θα επηρεάσουν ούτε αυτές αρνητικά τα υψηλά μας πρότυπα. Ε, ένα τρίτο πεδίο ωφελών, αυτό βέβαια το οικονομικό κέρδος. Η αξία είναι εξής, 4,7 εκατομμύρια ε, ε, θέσει εργασία στην Ευρώπη οφείλονται στι εξαγωγέ μα προ τι ΗΠΑ. Θέλουμε και άλλε εξαγωγικέ δυνατότητε και άλλη ζήτηση για, αυτούς, για αυτό το τι καλοπληρωμένε δουλειέ. Θέλουμε επίση το TTIP να ωφελήσει του καταναλωτέ, να έχουν μεγαλύτερη επιλογή σε χαμηλότερε τιμέ χαμηλότερες τιμές αγαθά και προϊόντα και υπηρεσίε. Ε, για τις εταιρείες μας επίσης. Οι εισαγωγές και τελικών προϊόντων και ενέργειας και πρώτων υλών θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Το 30% του συνολικού εμπορικού κύκλου εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τις εισαγωγές. Εδώ λοιπόν μπορούμε να φέρουμε πάλι πίσω ένα μέρος ευημερία στην Ευρώπη. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα για τις δημοσίες προμήθειες στη Φιλανδία. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται ΕΦΛΑ. Ε, η έδρα της είναι έξω από Φτιάχνουν εξοπλισμό για τα συστήματα φωτισμού που βοηθούν ε, τα αεροπλάνα αεροπλάνα να προσγειώνονται με ασφάλεια στου διαδρόμου των αεροδρομίων. Τα προϊόντα του έχουν εγκριθεί από τι Αμερικανικέ αρχέ, αλλά δεν μπορούν να του τα πουλήσουν, διότι ο Αμερικανικό νόμο δεν επιτρέπει παρά μόνο στι τοπικέ αρχέ να αγοράσουν εξοπλισμό εκτό ΗΠΑ. Εκτό και αν αυτό ο εξοπλισμό είναι άριστο. Ακόμη μάλλον και αν είναι άριστο. Ε, πρέπει όμω να είναι και προσαρμοσμένο σε πολύ δύσκολε καιρικέ συνθήκε. Όλοι θέλουν να αποφύγουμε τέτοιου είδου φραγμού. Για, για του δασμού στην Ισπανία. Διαφορετικέ εταιρείε έπρεπε να, να πληρώσουν πολύ ψηλού δασμού στι ΗΠΑ. Και πολλέ μικρομεσαίε στην παραγωγή τροφίμων, στα υποδήματα, έχουν ε, αναγκαστεί να πληρώσουν πολλού ε, δασμού. Στο Αλικάντε υπάρχει εταιρεία που πληρώνει 35% από το σύνολο του κόστου τη προ τι εκλογέ τη Αμερικανικέ. Και στην υπάρχει συγκριτικό μειονέκτημα με και προτιμούν να πολλούν προς τη Λατινική Αμερική. αλλά εκεί πληρώνουν 15% τέλη οι ευρωπαίοι επιχειρηματίε και εταιρείε. Επίσης υπάρχει μια μικρή εταιρεία που μια μικρή εταιρεία που παράγει ένα προϊόν από την πόλη που, από την οποία προέρχομαι το Smoothneck ε, που παράγει ένα μικρό ε, προϊόν το οποίο εξάγεται στι ΗΠΑ με δασμού 6%. Επίση, από το Τύρολο στην, στην Αυστρία ε, υπάρχει ε, εταιρεία που αναγκάζεται να υποστεί διπλό έλεγχο από τι ευρωπαϊκέ και τι αμερικανικέ για τη συμμόρφωση με του ίδιου κανόνε. Τα φάρμακα του γίνονται πολύ ακριβά για να απολύθουν στι ΗΠΑ. Και η Alfred Schuttingham, η οποία στην ε, κολονία, ε, στο, στην κολονία λοιπόν με τις παραγωγές ε, και πρίζας και άλλων προϊόντων ε, δεν καταφέρνει με 10-15% δασμούς να προωθήσει τα προϊόντα της στην Αμερικανική αγορά. Έπειτα στη Μεσογειακή ακτή της Γαλλίας, τα στρίβια. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την Αμερικανική αγορά γιατί δεν έχουν πια τα ρωσικά στρίβια. Αλλά δεν μπορούν να τα εξάγουν στις ΗΠΑ προς τη στιγμή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν διαφορετικού τρόπου ελέγχου των στριβιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάζει το ε, δίθυρο μαλάκιο το ίδιο, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, κοιτάζει το σύνολο. Κοιτάζουν το σύνολο. Το νερό. Οπότε Όλα αυτά είναι παραδείγματα για να αναγνωρίσουμε η μεν τα πρότυπα των δε τουλάχιστον. Θα εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χρήμα και πολύ χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του TTIP. Πραγματικά ε, χειροπιαστά ζητήματα για τι εταιρείε που σήμερα ήδη λειτουργούν και όλε αγωνίζονται σε μια οικονομία που χρειάζονται περισσότερε θέσει εργασία, περισσότερε επενδύσει και περισσότερο κέρδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευκαιρίε για τι μικρομεσαίε και τι μεγάλε εταιρείε. Ε, θα μπορούσαμε ε, να βελτιώσουμε τη λειτουργία των κυβερνήσεων μα με την τόνωση τη συνεργασία και να διαφυλάξουμε και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή που αλλάζει ούτω ή άλλω ταχύτητα και όπου υπάρχουν αξίε που δεν τι συμμερίζονται οι υπόλοιποι διεθνεί μα εταίροι. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε αν συνεργαστούμε. Σίγουρα αξίζει την ε, προσπάθεια και αναμένω να συνεχίσω τη συνεργασία μαζί σα με το Ευρωκοινοβούλιο και πολλού από εσά του εταίρου που είσαστε σήμερα εδώ για να επιτελεστεί πρόοδο αυτά τα ζητήματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση αυτή τη ακρόαση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε Μάλμστρομ, για τις αυτές αυτές δηλώσεις ε, Προ όφελο των πολιτών. Έχουμε εδώ 7 εκπροσώπους ε, των Ευρωπαίων πολιτών για να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Hm? Äh, Έχουμε τώρα 7 εκπροσώπους από διάφορες ε, ενώσεις των Ευρωπαίων πολιτών και θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις τους για την τύπα. Θα είναι κάπως διαφορετική η παρουσίαση από ό,τι ήθιστε στις ε, ακροάσεις. Θέλουμε να δώσουμε λίγη ζωντάνια. Θα είναι πολύ σύντομε λοιπόν οι εισαγωγέ και μετά θα έχουμε γύρω έρωτα απαντήσεων. Και ελπίζουμε και μια ζωντανή συζήτηση μετά τις 7 παρεμβάσεις και προκειμένου να είναι πραγματικά ζωντανή η συζήτηση και να λειτουργήσει με μεγάλη τεχνογνωσία, έχουμε εδώ την κυρία Βοντάν εδώ, η οποία είναι το πρόσωπο του EU Trade Insights, μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε κάποιες ε, περιπτώσεις να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι η κυρία Βοντάν ξέρει πολύ καλύτερα τι θέλουμε στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική από ότι και εγώ ο ίδιος. Είναι πολύ καλά λοιπόν ενημερωμένη και χαίρομαι ιδιαίτερω που βρίσκεται εδώ μαζί μα σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιωχάννα Κλάις από την ε, υπηρεσία BOIC, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ένωσης των Καταναλωτών. Και να σας πω επίσης ότι υπάρχει σχεδόν ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σήμερα στο πάνελ. σπάνια κι αυτό. Πέντε λεπτά λοιπόν ε, κατά το όριο. Ο κύριος Κλάης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα για τις ε, δυνατότητες που δίνει το TTIP για τους Ευρωπαίους και εκεί είμαστε ε, οργάνωση καταναλωτών, θα σας το παρουσιάσω υπό τη σκοπιά των καταναλωτών. Βέβαια το TTIP είναι ένα ευρύτατο θέμα, πολύπλευρο, ξεπερνάει τις ε, παραδοσιακές πτυχές του ανοίγματο αγοράς και της θεσμολογικής μείωσης. Το πιο προφανές ε, όφελος για μια εμπορική συμφωνία είναι φυσικά το οικονομικό. Ο πλούτος, η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών και εδώ κατά τη γνώμη μας υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί εμείς ως οργάνωση καταναλωτών δεν έχουμε τους πόρους και τη δυνατότητα να εκπονήσουμε διεξοδικές μελέτες επιπτώσεων. Αυτές ε, οι υπάρχουσες μέχρι τώρα μελέτες επιπτώσεων είναι αλληλονερούμενες. Οι αντίστοιχες μελέτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι 545 ευρώ ε, επιπλέον εισόδημα ε, για μια τετραμελή οικογένεια. Αυτό είναι αρκετά φιλόδοξη και αισιόδοξη ρυθμίση, ενώ άλλε μελέτε μιλούν για πιθανέ σημειέ στο ΑΕΠ ή απόλυε 0,50%. Βλέπετε, φάσκουν και αντιφάσκουν ακόμη και εμπειρογνώμονε. Δύσκολο λοιπόν μια οργάνωση καταναλωτών να, να διαμορφώσει γνώμη. Άλλωστε, οι δεσμολογικέ μειώσει είναι ένα μικρό τμήμα του TTIP και το άνοιγμα των αγορών. Είναι πολύ πιο πλευρή, πολύ πλευρή συμφωνία το TTIP. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να αποστοκοποιήσουμε τα ωφέλη και να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για, το, για την αύξηση του εισοδήματο ή τον πλούτο που θα δημιουργήσει μια τέτοια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ωφέλη, φυσικά μπορούμε να διδαχτούμε από εμπειρίε του παρελθόντο. Και εκεί φτάνουμε στα πιο προφανή θέματα. Άνοιγμα αγορών, δοσμολογικέ μειώσει και ανταγωνιστική πίεση στι αγορέ. Από αυτή την άποψη, το όφελος της TTIP είναι το πιο προφανές η μείωση των δεσμών γιατί οι δασμοί αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων, οπότε η μείωση των δασμών θα κάνουν τα προϊόντα πιο φτηνά, κάτι που ωφελεί τους καταναλωτές. Βέβαια, οι δασμοί είναι σχετικά χαμηλοί σε ό,τι αφορά το εμπόριο με τις ΗΠΑ, οπότε πόσο ακόμη θα χαμηλώσουν και τι όφελος θα έχουν τελικά οι καταναλωτές. Επίσης, επιλογή για τους καταναλωτές είναι ένα προφανές όφελος μιας εμπορικής συμφωνίας και της TTIP ότι διευρύνεται η επιλογή, το φάσμα των επιλογών. Αλλά θα πρέπει να δούμε εδώ ε, τις επιλογές ανατομέα για να δούμε πραγματικά τι κερδίζει ο καταναλωτής σε κάθε τομέα. Γιατί για ορισμένους τομεί μπορεί να διευρύνονται οι επιλογές, τα ψηφιακά προϊόντα, οι ψηφιακέ υπηρεσίε, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και σε μερικού τομείς όπου οι καταναλωτέ ενδιαφέρονται περισσότερο για ντόπια τοπικά προϊόντα, εκεί τα... οι επιλογέ δεν θα βελτιώνονται τόσο πολύ. Επίσης, ε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και στο παρελθόν, ε, με τις εμπορικές συμφωνίες, έχουμε νέες εισόδους στην αγορά, κάτι που αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση στους ε, διάφορους φορείς της αγοράς. Οι επιχειρήσεις κάνουν, μειώνουν τις τιμές για να έχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η είσοδος Ιαπωνέζικων και Κορεατικών αυτοκινήτων στην αγορά έχει φτηνίνει και τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Οπότε οι καταναλωτές ε, έχουν πρόσβαση σε φθηνότερα προϊόντα και σε μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Αυτό είναι φυσικά προς όφελός τους. Το θέμα είναι ότι ε, η TTIP δεν περιορίζεται στις δασμολογικές μειώσεις και στο άνοιγμα των αγορών. Γιατί από αυτή την άποψη υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές. Θα πρέπει όμως να δούμε και άλλα θέματα. Το πλαίσιο προστασία του καταναλωτή της Διατλαντικής Συμφωνίας για να κρίνουμε και από εκεί τα ωφέλη της TTIP. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, αν το TTIP ε, θέλει να είναι αποδοτικό, χρειάζεται μια ρωμαλαία πολιτική ανταγωνισμού. Γιατί ίσως τα εμπορικά ωφέλη εξουδετερωθούν από ε, απώλεια των ε, κερδών για τους καταναλωτές και όφελος μόνο των εμπόρων. Επίσης, για να κάνει ο καταναλωτή την καλύτερη επιλογή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεκμηριωμένη ενημέρωση. Επίση, θέλουμε ισχυρέ ρυθμιστικέ αρχέ που να μπορούν να δρουν ε, σε περίπτωση που εντοπίσουν ε, συμπεριφορά στρέβλωση στον ανταγωνισμού από τι εταιρείε. Επίση, δεν έχουμε μόνο το θέμα των καλύτερων τιμών. Θα πρέπει τα προϊόντα να είναι ασφαλή, να είναι υγιεινά και από αυτή την άποψη το θέμα της προστασίας, της ασφάλειας των προϊόντων ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και εκεί η σύγκριση, η μάλλον συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ε, είναι πολύ σημαντική. Να έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, κοινούς ελέγχους, ομοιόμορφα πρότυπα και προδιαγραφές και φυσικά να ευθυγραμμιστούμε με βάση τα πιο φιλόδοξα πρότυπα και τις ανώτερες προδιαγραφές και να μην έχουμε υποβάθμιση των προδιαγραφών. Μετά από διετής διαπραγματεύσεις ε, δεν μπορούμε να πούμε αν η προσέγγιση αυτή τη σύσταση ενός ε, πλαισίου προστασίας του καταναλωτή που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αυτά. Θα είχα και άλλα πολλά να σας πω, αλλά προτιμώ να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ, Ιωάννης. Μιλήσατε για υψηλά πρότυπα. Αυτό είναι πολύ α, φυσιολογικό για τους καταναλωτές. Όλοι θέλουμε υψηλά τα πρότυπα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο υψηλά τα πρότυπα στις ΗΠΑ και όχι στην Αμερική και όχι στην Ευρώπη. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι το TTIP είναι η πιο σωστή μορφή εννοπής, ενσωμάτωση των ε, αμερικανικών προτύπων. Μήπω πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα και ίσω το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να σκεφτεί κατάρτιση δικιά μα νομοθεσία πρώτου την εντάξουμε στο TTIP η απάντηση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Καταρχά υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν ε, έχουν να κάνουν μόνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πλέον, κοιτώντα για παράδειγμα περισσότερο εμπόριο στα τρόφιμα, στα χημικά, στα ε, καλλιτικά. Δεν πρέπει, δεν μπορούμε να υπολογίζουμε μόνο σε υψηλά πρότυπα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από άλλες αγορές που δεν πληρούν τα πρότυπά μας. Η Επίτροπος Μάλμστρομ μίλησε πριν από λίγο για τα ανανοηλικά και την ενδεχόμενη συνεργασία στον τομέα αυτό. Από την αρχή των διαπραγματεύσεων Έχουμε ακούσει διάφορες προτάσεις για θετικά ζητήματα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, τα οποία θα πρέπει να δεκτάξουμε με την ΕΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα ανηλικά, για παράδειγμα, γιατί να μην συζητάμε με τι ΕΠΑ το πώς μπορούμε να συστήσουμε ένα σύστημα μητρώου για τα νοηλικά, το στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι νομοθέτες αλλά και το ευρύ κοινό. Γιατί να μην κάνουμε μια αξιολόγηση πριν από την εμπορία των ανών υλικών προτού επιτρέψουμε την διάθεση στην αγορά καλλιντικών ή χημικών. Και το ίδιο ισχύει και για άλλους τομείς, όπως το τρόφιμα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου καλό θα ήταν να σκεφτούμε το εμπόριο με τις ΙΠΑ, αλλά με τον πιο υψηλό κοινό παρανομαστή πάντα ως βάση. Και στο αυτό μπορεί να έχει νόημα. Γιατί αν υπάρξει πιο πολύ εμπόριο στα τρόφιμα, θα πρέπει να εξετάσουμε δύο πιο παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγή γιατί στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει κίνδυνο να εισαχθούν στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα. Όταν μιλάμε δηλαδή για το TTIP θα πρέπει να μιλάμε παράλληλα για ένα νέο σύστημα ανεκνευσιμότητα μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να εντοπιστεί ο παραγωγός ή κάποιο παγκοσμίο σύστημα ειδοποίησης αν εισαχθούν προϊόντα από τις ΙΠΑ, η τρόφιμα για παράδειγμα πάλι και στην Καλιφόρνια ο κόσμος ε, ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά με τα πορτοκάλια για παράδειγμα να μπορούν να ενημερωθούν οι αρχές ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο γρήγορα. Ναι, μία επερώτηση. Θα επιμένω εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει εδώ και καιρό ότι το ΔΤΠ δεν πρόκειται να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Φυσικά αυτό το λένε σε ό,τι αφορά όλες τις ανησυχίες για τη μείωση των προτύπων μας. Αλλά το ίδιο δεν θα είναι, δεν θα ισχύει. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τα πρότυπά μας, δεν είναι λίγο αφελές από πλευράς της Ένωσης Καταναλωτών. Και συγγνώμη αν κάνω κριτική να θεωρούμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα του TTIP. Αν θέλετε να μου απαντήσετε στην συντομία, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο είναι η απάντηση. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο. Πρωτού ξεκινήσουμε πιο εκτεταμένε εμπορικέ σχέσει με τι ΗΠΑ και με άλλου εταίρου, να σκεφτούμε και κάποιου από του κινδύνου που συνεπάγεται αυτή η εμπορική σχέση για μεγαλύτερο, εμπόριο, για παράδειγμα, σε αφορά τα χημικά, τα καλλιτικά. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο κάποιων προϊόντων που παράγονται με τρόπο που δεν πληρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό λοιπόν, είτε μέσω του DTIP είτε μέσω άλλων πλατφόρμων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο, η Φαμπιέν Φωνίσλαν, η οποία εργάζεται για την καλλική εταιρεία παραγωγής ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ονομάζομαι Φαμπιέν Γκογιανές και θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα το τι μπορεί να προσφέρει σε έναν όμιλο όπως η Μισλά μια συμφωνία σαν το TTIP. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω κάποια στοιχεία για την ε, Μισλά που εξηγούν τις προσδοκίες μας. Αν έρθατε σε αυτήν την ε, ακρόαση με το ποδήλατο, το μετρό ή το αεροπλάνο ή το λεωφόριο ε, μπορεί, ή το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιήσετε μισελέν χωρίς να το γνωρίζετε γιατί πρόκειται για ε, λάστιχα που ε, τα παράγουμε εμείς. Μαύρα, απλά, αλλά με μια, ένα συμπίκνωμα τεχνολογίας. Μέχρι και 200 συστατικά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν. Αυτό φυσικά έχει τεράστιο αντίκτυπο ως προς το διεθνές εμπόριο για μας. Ε, ε, η Μισλά είναι μια εταιρεία ε, διεθνής. Έχει εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, 37 εργοστάσια παραγωγής, ένα κέντρο έρευνας και 60.000 εργαζομένους. Του μισού εργαζομένου του ομίλου και 60% τη παραγωγή του ομίλου σε τόνου. Επίσης έχουμε κατασταθεί εδώ και πολύ καιρό στις ΗΠΑ διότι έχουμε εργαστάσει από το 1975 με στόχο να καλύψουμε την Αμερικανική αγορά. Σήμερα έχουμε 16 εργοστάσια και ένα κέντρο έρευνα και παραγωγή και πάνω από 18.000 εργαζομένου. Ε, για μα το TTIP έχει ε, πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για τη Μισλά. Έτσι κι αλλιώ, εμεί έχουμε ισχυρή παρουσία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με ένα προϊόν που είναι περίπλοκο και αποκρίνεται σε διάφορες ειδικές ανάγκες. Έτσι, έχουμε ροές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σημαντικές, και αυτό που αναμένουμε από το TTIP είναι κυρίως κέρδος ως προς την παραγωγικότητά μας, ε, με την κατάργηση των τελωνιακών δεσμών που τόσο άλλως υπάρχουν και από τις δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Ε, ε, πρέπει να πούμε ότι οι δασμοί των, το ύψος των δασμών είναι γύρω στο 3% για το, τα αλλά 6% για τα χημικά προϊόντα. Οι ροές όμως είναι πολύ υψηλέ. 37% της ευρωπαϊκής παραγωγής εξάγεται και το 40% προς τι ΗΠΑ. Οι ροές είναι πολύ σημαντικέ λοιπόν και αυτό επηρεάζει την αγορά. Εάν σκεφτούμε τα λάστιχα ε, για τα φορτηγάκια. Συνήθω αυτά τα παράγουν Ευρωπαίοι παραγωγοί. Στην Ευρώπη, όταν πρέπει να καλύψουμε με τέτοια λάστιχα τι ΗΠΑ, τα εξάγουμε από τα ευρωπαϊκά μα εργοστάσια. Αντιστρόφω, για τα 4x4, που είναι ένα ε, εργοστάσιο εξοχήν αμερικανικό, έχουμε εργοστάσιο εκεί που παράγει λάστιχα για τα τζιπ. Ε, όταν πρέπει λοιπόν να παράγουμε τέτοια λάστιχα, τα φέρνουμε ε, και στην Ευρώπη από τι ΗΠΑ. Τώρα, για τα λάστιχα του μετρό. Θα το έχετε δει σε μετρό από τα αεροδρόμιο. Αν πάτε στην Disneyland, στο Νέα Υόρκη, στο Μαϊάμι και ούτω καθεξή. Αυτά τα ελάχιστα παράγονται ε, αποκλειστικώ στην Ευρώπη, κατευθύνονται προ την Ευρώπη και έχουν 3% ε, δασμού τελωνιακού στην είσοδο προ τι ΗΠΑ. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει ότι οι τελωνιακοί δασμοί μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την επιχείρησή μα, αλλά και άλλου ομίλου ε, από, το, από την κατά συνεπτοχικά είναι κάτι που είναι τα, ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μηχανήματα με δασμούς, τελωνιακούς δασμούς 6%. Εάν μειώσουμε αυτούς τους τελωνιακούς δασμούς, αυτό θα ωφελούσε και εμάς και όλη την αλυσίδα παραγωγής μηχανημάτων στην Ευρώπη. Ως προς τους αριθμούς, οι ροέ αυτέ, των οποίων σα έδωσα κάποια παραδείγματα, εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίω για να όμιλο στον δικό μα. Αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ ελπίζουμε ότι θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν να κάνουμε το μηχανικό μα και παραγωγικό μα εργαλείο στην Ευρώπη πιο αποτελεσματικό. Κάπω λίγο πιο ανταγωνιστικό και έτσι θα μπορούσαμε να δούμε το TTIP ως ευκαιρία πλούστευσης των διαδικασιών, καταργώντας κάποιους φόρους ε, στους οποίους πρέπει να υποκληθούμε σήμερα. Λόγω χάρη κατά την είσοδο στις ΗΠΑ υπάρχει ένας φόρος που ονομάζεται σε ωραία γαλλικά Merchandise Processing Fee. Αυτό θα πει ότι για κάθε εμπόρευμα, κάθε παρτίδα που εισάγεται πληρώνουμε 500 ε, δολάρια. Με τη συμφωνία ναύτα και ε, με το TTIP επιτέλους κάποια στιγμή θα μπορούσε αυτός ο δασμός να εξαλειφθεί. Ε, συμπερασματικά λοιπόν η συμφωνία TTIP για να όμιλο το δικό μας θα προετρέψει να κερδώσει την παραγωγικότητα που θα το επιτύχουμε με την κατάργηση των κλινικών δασμών. Έχουμε ροές πολύ σημαντικές μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Μιλούσα για ροές προϊόντων αλλά θα μπορούσα να μιλήσω και για ροές ανθρώπων ανδρών και γυναικών. Έχουμε μετανάστες από τι ΗΠΑ στην Ευρώπη και μετανάστες από την Ευρώπη στι ΗΠΑ. Αν δεν αντιμετωπίσουμε του ελληνικού δασμού σήμερα, πιστεύουμε ότι θα χάσουμε μια μόχλευση ανταγωνιστικότητα με το TTIP, γιατί θα μπορούσαμε πραγματικά να τι εξαλείψουμε αυτέ τι βιομηχανικέ δυσκολίε. Ε, το βιομηχανικό μα εργαλείο στην Ευρώπη, που έχει εξαγωγικέ ε, τάσει, να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό στο διεθνέ προσκήνιο, με τα πλαίσια τη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, Φαμπιέν. Ε, εξεπλάγην κάπω. Μιλήσατε πάρα πολύ για πλήρη εξάλληψη των ε, τελωνιακών δασμών. Και είπατε ότι υπάρχουν και πολλοί Αμερικανοί που είναι εδώ. Και αντιστρόφω, φαντάζομαι το ίδιο και με του εμπειρογνώμονε. Θα ταξιδεύουν και από τη μια και από την άλλη. Και θα υπάρχουν και κέντρα στι ΗΠΑ που έχουν ανάγκη από πληροφοριών. Δεν υπάρχουν φραγμοί σε, σε αυτέ τι κατηγορίε. Μόνο στου ελληνικού δεσμού έχετε πρόβλημα. Κοιτάξτε, μιλάω περισσότερο για ρυθμιστική σύγκληση μάλλον. Ε, αυτό εννοώ. Έχετε δίκιο το αμερικανικό σύστημα και το ευρωπαϊκό σύστημα για τα λάστιχα είναι τελείως διαφορετικά. Ε, δεν ε, λειτουργούν τον ίδιο τρόπο. Έχουμε διαφορετική έγκριση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Έχουμε όμως παρουσία 40 χρόνων στις ΗΠΑ έχουμε έναν τρόπο να, έχουμε έναν τρόπο να αντιμετωπίζουν το θέμα που εμείς το έχουμε καλύψει πλήρως πλέον. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό για μας και να πω και τα εξή. Από τη μια, εάν το TTIP μπορούσε να είναι μοχλός για τους φορείς όπως αυτός της Γενέβης, τον ΠΟΕ, για να περάσουμε σε μεγαλύτερη αναρμόνιση των ε, συστημάτων μας, αυτό θα ήταν ήδη ένα ενδιαφέρον θέμα για μας και στο μέλλον, και μετά αυτό που θα μπορούσε να μας φανεί ενδιαφέρον είναι οι χρήστε των χημικών προϊόντων. Ο ρυθμιστικό διάλογο θα μπορούσε να προκύψει μέσα από τη συμφωνία TTIP μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να μα ενδιαφέρει να δούμε πώ θα έχουμε πιο καλέ, πιο έντονε ανταλλαγέ για το θέμα των χημικών προϊόντων, λόγου χάρη. Ε, ναι, αλλά να κάνω και περώτηση. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο τα χημικά προϊόντα. Μιλάμε πολύ για τον κίνδυνο απορρίθμιση από την οδηγία REACH Οπότε παρακαλώ να είστε απόλυτα ειλικρινεί. Θα είναι κάτι που θα σα ωφελήσει, εάν ανακριθεί η REACH. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό ο στόχο τη συμφωνία TTIP. Η συμφωνία REACH έχει επιτρέψει σημαντική πρόοδο σε όλου του τομεί και ω προ τη διαφάνεια και για χρήστε όπω εμεί και επειδή είναι ο τελικό μα στόχο ω προ την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Καθόλου δεν επιθυμούμε την ε, εξάλληψη της οδηγίας REACH. Ο τελικός στόχος του REACH είναι να λειτουργήσει ως μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μέσω του ελέγχου των χημικών συστατικών, των χημικών ουσιών. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει με το TTIP είναι ότι εφόσον κάθε γεωγραφική περιοχή θα έχει το δικό της, έχει μάλλον τώρα το δικό της σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση το REACH και η Αμερικανοί άλλο σύστημα, στο διάλογο μας ε, εκ των, προτέρων, προφανώς αν μια ουσία κρίνεται επί βλαβερή στην Ευρώπη θα είναι βλαβερή και για, για τους Αμερικανούς. Οπότε ο τρόπος που κάνουμε την επιστημονική μας αξιολόγηση των ουσιών που ε, ε, προσπαθούμε να τις κάνουμε λιγότερο βλαβερές, θα μας αναγκάσει να έχουμε εντονότερο διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη προβλέψιμότητα για το δικό μας εμπορικό κλάδο και αυτό θα είναι πιο ενδιαφέρον και για τους πολίτες από την άποψη της υγείας και του περιβάλλοντος. Εάν αυτός ο διάλογος είναι πιο εντατικός ε, νωρίτερα από την εμπορματοποίηση. Ονομάζεται RIT και είναι νομοθεσία στην Ευρώπη, έχει άλλο όνομα στις ΗΠΑ, αλλά ο τελικός στόχος είναι ο ίδιος. Είπατε ότι τα τελωνιακά, ε, ελληνική δασμή είναι 20 εκατομμύρια ετησίω. Α φανταστούμε ότι καταργούνται πλήρω οι ελληνική δασμή. Κερδίζετε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα κερδίσω εγώ. Συγκεκριμένα, τι θα τα κάνουμε τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ερώτησή σα, μάλλον δύσκολο να σας απαντήσω έτσι, γιατί η αγορά των ε, λάστιχων είναι πολύ ανταγωνιστική ε, και εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Αν σας έδινα αριθμούς το 2000, η 10 πρώτη παραγωγή λαστίχων στον κόσμο ήταν περίπου 80% το μεριδίου της αγοράς. Το 2013 η 10 πρώτη παραγωγή λαστίχων στον κόσμο φτάνουν το 60% της παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια χάσανε 20% του μεριδίου αγοράς λόγω της ανάδεσης νέων συμμετεχόντων στην αγορά. Τεράστιος ανταγωνισμός. Σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά του λάστιχου δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που γνώριζαμε πριν την κρίση. Εάν δούμε αυτή την εξέλιξη που είναι τόσο γοργή, ε, αυτή η διεθνής αγορά που είναι τόσο ανταγωνιστική, Είναι πολύ δύσκολο να σα πω τη στιγμή που το TTIP θα εγκρινόταν, θα κυρωνόταν και θα υλοποιητό, τι θα το κάναμε ε, αυτό το 20 εκατομμύρια που θα κερδίζαμε. Να θα το αξιοποιούσαμε για την ανταγωνιστικότητα, για να εξοχρονίσουμε τα εργοστάσια και τη βιομηχανία μα στην Ευρώπη, για να καταρτήσουμε του εργαζομένου μα, για να συνεχίσουμε την έρευνα και την ε, ανάπτυξη προϊόντων. Δύσκολο να σας πω. Ε, όταν όλα αυτά μπορεί κάποτε να λάβουν χώρα, πού θα βρισκόμαστε είναι δύσκολο να το προβλέψω, Ελπίζοντα ότι οι διαπραγματεύσει θα προχωρήσουν γρήγορα. Σα ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά ελπίζουμε οι επενδύσει να είναι στην Ευρώπη. Ο κύριο Τίλμαν Κούπφερ από την British Telecom είναι ο επόμενο ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και από την British Telecom για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Αμερικανική αγορά για μας. Γι' αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το TTIP και πριν από 30 χρόνια ξεκινήσαμε και ανοίξαμε την πρώτη μας ε, εταιρεία στη Νέα Υόρκη όταν είχαμε μπει και στο αμερικανικό χρηματιστήριο τότε που είχε ιδιωτικοποιηθεί η BT, British Telecoms. Έκτοτε έχουμε ανοίξει και άλλα γραφεία στο Χιούστον και σε πολλές άλλες πόλεις. Ε, δυνάτη Σαν Χωσέ και το καθεξής. Και έχουμε ε, 2.200 εργαζομένους στις ΕΠΑ. Είναι η πιο σημαντική λοιπόν εθνική αγορά η ΕΠΑ εκτός από την, το Ρεμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν μια φιλόδοξη συμφωνία TTIP για μας για να υπάρχει αμοιβαίο όφελο. Έχουμε επίσης υποστηρίξει και άλλες πολυμερείς και διμερείς εμπορικές διαδικασίες διαπραγματεύσεις τις οποίες ε, κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά, την Κορέα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρ, την Μερκοσούρ και το καθεξή. Είμαστε ο μεγαλύτερο πάροχο ε, ε, σταθερών επικοινωνιών στην Ηνωμένη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και λειτουργούμε σε 170 χώρε. Και εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου δεν παρέχουμε υπηρεσίε σε ε, ιδιώτε, αλλά σε επιχειρήσει, μεγάλε, μικρέ επιχειρήσει, μικροεπιστήμες επιχειρήσει που λειτουργούν στο διεθνές προσκήνιο, κυβερνήσει, διεθνού οργανισμού κτλ. Έχουμε παγκόσμια παρουσία που συνδέει όλες τις μεγάλες πόλεις στον κόσμο και επενδύουμε σημαντικά ποσά στην έρευνα και στην ανάπτυξη για την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων σε θέματα ICT για να ανταποκριθούμε στις ανάγκε των πελατών μας. Άρα αυτό ήθελα να σα το λέω να σα καταδείξω ότι δεν περιοριζόμαστε στις κλασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Και φυσικά πιστεύουμε στην BT ότι το εμπόριο σχετίζεται ε, με την μεγαλύτερη χρήση των ε, υπηρεσιών ICT και αυτό δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε επίσης πρόσβαση στις ε, πολιτιακές διαδικασίες παροχής συμβάσεων διαγωνισμών στις ΕΠΑ και πιστεύουμε ότι χρειάζεται ελεύθερη ροή δεδομένων με την, για την καλή λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών σε όλους τους τομείς και αυτό θα πρέπει να συνάδει με μια φυσικά ισόρροπη προστασία των δικαιωμάτων έθεν και έθεν του αφαντικού. Προσβλέπουμε σε μια φιλόδοξη συνεργασία για θέματα κανονιστικά για να αντιμετωπίσουν το θέμα των νέων υπηρεσιών και των μελλοντικών προτύπων που θα πρέπει να ισχύουν σε νέους τομείς όπως είναι η ηλεκτρονική υγεία, το νέφος ε, και τέλος θέλουμε μια συνεκτική προσέγγιση στην, ε, στους κανονισμούς στην νομοθεσία που αφορούν την πρόσβαση στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Για το τελευταίο αυτό σημείο πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία μας ε, θέλει στα πλαίσια της συμφωνία του TTIP να αντιμετωπιστεί το θέμα των εμπορικών φραγμών και αυτό περιλαμβάνει τα θέματα ειδική ε, πρόσβασης όπως αναφέρονται στο, στη ΣΥΠΑ. Στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών τα εμπορικά προσκόμματα κατηγοροποιούνται σε τρεις κατηγορίες. Καταρχά έχουμε την έλλειψη απελευθέρωση όπου δεν έχουμε πρόσβαση. Έχουμε τα ανώτατα όρια αλλοδαπών επενδύσεων, όπου έχουμε περιορισμένη δηλαδή πρόσβαση. Και τέλος έχουμε ε, προβληματικές ε, νομοθεσίες και κανονισμούς για την διαχείριση των αγορών, όπου υπάρχει δηλαδή πρόσβαση αλλά με προβλήματα. Και θεωρούμε ότι στο τελευταίο τομέα ε, είναι εκεί που εστιάζονται τα προβλήματα με τις ΕΠΑ. Οι μελέτες ε, καταδεικνύουν ε, τεράστια ωφέλη για τις τηλεπικοινωνίες από το TTIP. Από το 2013 ε, εντοπίζεται ότι θα μπορούσε να έχει όφελος από 19 δισεκατομμύρια ευρώ εάν υπήρχε καλύτερη ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ήδη υπάρχουν μεγάλα ωφέλη. Η μελέτη της αμερικανικής αγοράς που δεν ρυθμίζεται σωστά υπολογίζει 160 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα αυτό είναι αποφελές όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους καταναλωτές της ΕΠΑ. ΕΕ. Θα ήθελα κλείνοντα χωρί να επαναλάβω και από αυτά που είπε η κυρία Μάλμστρομ, θα ήθελα να πω το εξή. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια σχετική έρευνα για τα ωφέλη της ε, πρόσβασης ε, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και αυτό ασφαλώς αφορά πολλές ε, πόλεις και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Πραγματικές ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσατε για ελεύθερη ροή δεδομένων. Πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Και το σχέδιο ψηφίσματος του κ. Λάγκη για το DTIP θέλει να αποφευθεί οποιαδήποτε δέσμευση για ανταλλαγή δεδομένων πριν ε, ε, τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πώ μπορείτε να τον πείσετε περί του αντιθέτου. Όταν μίλησα για ροή δεδομένων, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνεται με βάση τους ε, υπάρχοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Αλλά υπάρχουν και άλλες ανησυχίες, αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις για παράδειγμα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και πέραν της ε, προστασίας δεδομένων καθ' αυτής στο TTIP. Γιατί γίνονται εκ παραλλήλου και άλλες ε, συνομιλίες και διαπραγματεύσεις. Οπότε χρήσιμο θα ήταν αυτές οι παράλληλες συζητήσει ε, να προχωρήσουν για να ολοκληρωθεί έγκαιρα και η TTIP. Δηλαδή συμφωνείτε να μην υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στο TTIP για την προστασία των δεδομένων. Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ανησυχίε και προ το παρόν δεν θέλετε ένα τέτοιο ειδικό κεφάλαιο στην TTIP. Εντάξει, μπορεί να φανώ κακή, αλλά η British Telecom ήταν στο επίκεντρο ενό σκανδάλου για την προστασία των δεδομένων και την προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Γιατί τώρα το προωθείτε και μάλιστα εντός της συμφωνίας TTIP. όπως είπα, αφορά τις δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων, ε, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Δεν είναι μόνο δικό μας, ε, δικός μας προβληματισμός και μέρημνα. Εγώ αναφέρθηκα στη, στις, ένα, σε ένα ισχυρό κεφάλαιο για, για τις υπηρεσίες αυτές για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση ε, των τηλεπικοινωνιών. Ναι, το καταλαβαίνω συνεργάστηκε με την Επιτροπή τώρα. Για τι δημόσιε συμβάσει. Τεράστιο θέμα. Εκεί έχουμε ομοσπονδιακό σύστημα στι ΗΠΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μάχη του επόμενου μήνε για να συμφωνήσει σε ένα επίπεδο δημοσίων συμβάσεων, ένα πολιτιακό επίπεδο, όχι ομοσπονδιακό δημοσίων συμβάσεων. Αν δεν έχετε τέτοιο υπό-ομοσπονδιακό, δηλαδή πολιτιακό ε, σύστημα δημοσίων επενδε... συμβάσεων. Ποια θα είναι η επίπτωση για σας. Φυσικά θα δημιουργηθούν ε, περισσότερες επιχειρησιακές ευκαιρίες, ε, περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να ανοίξει το πολιτιακό επίπεδο δημοσίων συμβάσεων, να μην γίνονται όλα δηλαδή σε κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Και το άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων είναι ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο το που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε καλύτερη ανταγωνιστική θέση στην Αμερικανική αγορά. Και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι άλλοι εμπορικοί φραγμοί πλην των δασμών. Η ΕΠΑ έχει παρόμοιες διατάξεις με άλλες χώρες του ΩΣΑ. Αλλά διαφέρει από τη η Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάζομαι ότι για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας θέλετε μια ζωντανή συμφωνία. Και φαντάζομαι θα είναι υποχρεωτική για σας αν θέλετε να συμμετέχετε στη συμφωνία και να αποκομίσετε και καρπούς και ωφέλη από τη συμφωνία. Αναφέρθηκα στη της μυστική μη κανονιστική συνεργασία για τις υπηρεσίες, νέες υπηρεσίες σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Σίγουρα αυτό θα ήταν το ζωντανό τμήμα της συμφωνίας. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Περνάμε στην άλλη όψη του νομίσματος, στα συνδικάτα και στην κυρία Σουζάν Λίμπερκ, που εκπροσωπεί τη Σουηδική Ομοσπονδία Συνδικάτων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Θα σας παρουσιάσω και κάποιες διαφάνειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεπεράσω τα πεντά λεπτά που μου δώσατε. Πάντως χαίρομαι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ω Ευρωπαίο πολίτη που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι γιατί αξιοποιούμε το δημοκρατικό πλεονέκτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορούμε να μιλήσουμε και τη μητρική μα γλώσσα όλοι. Γι' αυτό θα αξιοποιήσω αυτό το πλεονέκτημα το δημοκρατικό. Όσοι δεν γνωρίζουν τη Σουηδική παρακαλώ να φορέσουν τα ακουστικά του. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να σα μιλήσω σήμερα για την συνδικαλιστική σκοπιά του TTIP. Τι θα κερδίσουν οι Ευρωπαίοι από την διατλαντική Ευθυντερική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Οι διαφάνειες που έχω ετοιμάσει είναι στα αγγλικά, αλλά εγώ θα μιλήσω σου Ελπίζω να βλέπετε καλά την ε, οθόνη ταξιδικά συνδικάτα πριν από ένα χρόνο ενέκριναν ένα πολιτικό έγγραφο για το TTIP. Οι τρεις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις της Σουηδίας ε, εκπροσωπούν 70 ε, με 80% των Σουηδών εργαζομένων. Η Σουηδία είναι χώρα εξαγωγές. Εξαρτάται λοιπόν από τις εξαγωγές της για να διαθέσει τα προϊόντα της. Και φυσικά Έχουμε μια πολύ θετική διάσταση απέναντι σε ελεύθερες συναλλαγές, γιατί ε, εκποιώντας, διαθέτοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας, ε, δημιουργήσαμε μια κοινωνία ευμάρειας με υψηλή φορολογία, βέβαια, στη Σουηδία. Οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες είναι επίσης ε, ευνοϊκές απέναντι στις ιδέες των ελεύθερων συναλλαγών. Τώρα, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους ε, εργαζόμενους. Πιστεύω ότι ένας θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ καλοπροαίρετων επιχειρήσεων και έντιμων θα είναι θετική για τους εργαζόμενους γιατί θα οδηγήσει σε υψηλούς μισθούς. Ναι, μεν, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η αγορά εργασία να είναι δεκτική απέναντι στι αλλαγέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική διαχείριση τη ανεργία και μια ε, πολιτική οργάνωση ε, τη αγορά εργασία που να είναι θετική απέναντι στι ε, ελεύθερε συναλλαγέ. γιατί θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από τη διατλαντική αυτή συμφωνία. Και το ελεύθερο εμπόριο, οι ελεύθερε συναλλαγέ προποθέτουν αντι... αντιστάθμιση των ζημιών από τα κέρδη. Γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Εμείς κρίναμε ότι συνολικά το TTIP έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα. Παρόλο που δεν συμμερίζονται όλε οι ισουηδικέ Συνδικαλιστικέ Οργανώσει το δικό μα ενθουσιασμό και αισιοδοξία για το TTIP. Περνάω στην επόμενη διαφάνεια. Πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Έχουμε 24 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρώπη. Βέβαια δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργία το DTIP, σίγουρα. Έχουμε τις ευρωπαϊκές δράσεις και τις εθνικές δράσεις που θα πρέπει να συμβάλλουν για τη διόρθωση του προβλήματο, αλλά και το DTIP θα βάλει το λιθαράκι του στη βελτίωση τη κατάσταση. Επίσης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Με το TTIP οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά. Και πιστεύουμε ότι σε περίπτωση διαφορών θα μπορούσε το πρόβλημα να διαθετηθεί σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θεωρούμε ότι από κοινού οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση παγκοσμιοποιημένων εμπορικών κανόνων. Είμαστε δύο δημοκρατικές κοινότητες που εστερνίζονται κοινέ αξίες και θέλουμε, θα θέλαμε αυτές τις δημοκρατικές αξίες να τις μεταλαμβαδεύσουμε και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Τώρα, είναι θετικό το TTIP για τους εργαζόμενους και υπό ποιου όρους. Είναι φυσικά σημαντικό να προασπίσουμε και να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των μισθωτών και των εργαζομένων. Βέβαια δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως εμπόδιο. Και το TTIP θα πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή των συμβάσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας Επίσης, ε, κάθε χώρα θα πρέπει να διασφαλίσει ένα περιθώριο λιγμών. Και το, τα εθνικά συστήματα ευμάρειας και κοινωνικής πρόνοιας δεν θα πρέπει να διακυβεύονται από το τι ούτε να υπονομεύονται από αυτό. Επίσης, η οδηγία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις ε, και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λαμβάνουν χώρα εύρυθμα και πρόσκοπτα. Ούτε είμαστε υπέρ του ISDS δεν είναι απαραίτητο αυτός ο μηχανισμός επίλυση διαφορών επένδυτου του κράτους. Θεωρούμε ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους πάντα στο TTIP, σε τελική ανάλυση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Είδα στην παρουσίαση PowerPoint ότι μιλήσατε για το μηχανισμό ISDS. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τρία πάνε να αναφέρουμε το ISDS. Θα ήταν μαγικό αυτό. Οπότε τι είπατε, να το δεχτούμε ή ότι πρέπει απλώς να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Στην... Ε, με συγχωρείτε. Καλά, εντάξει. Θα τα πω τώρα. Είπαμε ότι λέμε όχι στο ISDS. Διότι τα υπέρ και τα κατά δεν είναι παρόμοια. Η διαφάνεια, η δημοκρατική λογοδοσία και άλλοι λόγοι μας οδηγούν να λέμε όχι στα ISDS. Δεν είναι απαραίτητο σε μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ. Ωστόσο, εάν το ISDS υπάρξει συμπεριληφθεί στο TTIP και το παρακολουθήσουμε σωστά, θα δούμε ότι οι κανόνες που περιλαμβάνονται δυστυχώς στην συμφωνία με τον Καναδά ε, δεν είναι αρκετοί και όπως είπε και η Επίτροπος Μάστρομ θα υπάρξει τώρα ε, βελτίωση θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επηρεάσουμε και μέσω της κυβέρνησής μας και με άλλες ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις και το να μιλούμε για τα δικαιώματα των επενδυτών είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τις ευθύνες των επενδυτών ταυτόχρονα. Και πιστεύω ότι το θέμα πρέπει να το δούμε και με άλλους συναδέλφους από, από τον κόσμο των εταιριών. Να δούμε τι ακριβώ θέλουμε να ρυθμιστεί. Το δικαίωμα το ρυθμίζουν. Αλλά να οριστεί και στο διεθνέ εμπόριο η ευθύνη του επενδυτή και στι διεθνεί επενδύσει. Πώ έβεται κανεί τι κατευθυντήρε γραμμέ του ΠΟΕ για τι πολυεθνικέ και πώ και του ΟΣΕ και πώ τι αντίστοιχε αμερικανικέ. Αυτό είναι ένα ενιαίο πακέτο. Και ένα τρόπο για να λύσουμε το πρόβλημα του SDS είναι να έχουμε ένα βιώσιμο TTIP, αλλά και ένα συνολικό πακέτο για τι ευθύνε των επιχειρήσεων. Είπατε και για ψηλά εργασιακά πρότυπα. πώ, όχι εμεί, όχι εγώ, δεν δεν κάνω κάτι τίποτα, η Επιτροπή πώ μπορεί να διαπραγματευτεί το TTIP με έναν εταίρο που δεν έχει κυρώσει τι περισσότερε από τι συμβάσει του ILO, του, του Παγκόσμιου Οργανισμού εργασία και εφαρμόζει άλλα πρότυπα. Δεν σα ανησυχεί αυτό. Ναι, συζητήσαμε στη Στοκχόλμη τον Υπουργό για τα θέματα αυτά και το, το θέσαμε. Πώς μπορεί να υπάρξει σωστή επιβολή του κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Με, τα, με χαρά βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θέλουν ένα δεσμευτικό υποχρεωτικό κεφάλαιο με τα καλύτερα από την Αμερικανική πλευρά την οικονομική αιρεσιμότητα και τα καλύτερα από την ευρωπαϊκή πλευρά. Τα κείμενα, το περιεχόμενο. Ελπίζω και είμαι πεπισμένη. Ελπίζω τέλο πάντων ότι το TTIP θα κάνει νέα βήματα. Ω προ τι βασικέ συμβάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία. Ανυπομονούμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κυρώσουν καμιά από τι συμβάσει του ILO σας το είπε αυτό ο Υπουργός. Ε, όχι, θα ζητήσουμε όμως την κύρωση των βασικών συμβάσεων του ΕΛΟ. Αυτό το θεωρούμε απαραίτητη προπόθεση. Αλλά είπαμε κιόλα ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαιτήσει και αποτελεσματική υλοποίηση των συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Πραγματικά με πάρα πολύ από μια συνδικαλιστική οργάνωση. Βέβαια ξέρω ότι είστε από τη Σουηδία, είστε πιο φιλελεύθεροι από άλλε χώρε. Στη Γαλλία μια συνδικαλιστική οργάνωση θα είχε αντιδράσει τελείω διαφορετικά στην μη κύρωση των συμβάσεων του ΑΕΛΟ από τι ΗΠΑ. Τι λένε οι ομολογοί σα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τι πιστεύετε ότι θα προκύψει. Συζητούμε. Και βεβαίω συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και έχουμε διοργανώσει σεμινάριο από κοινού μαζί του στην Washington με την αντίστοιχη επίση Αμερικανική Συνομοσπονδία και είδαμε πώ θα αλλάξει η αγορά εργασία και πώς μπορούμε να ζητήσουμε κοινέ λύσεις ή να γίνει σωστή κατανομή με την ε, διάσταση της παγκοσμιοποίηση. Όμως, είναι σαφές ω προ το δικαίωμα, το απεργή και άλλα ζητήματα. Πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασία. Αλλά ω ε, πρώτο πράγμα θα πρέπει να έχουμε την κυρίωση των συμβάσεων του ΑΕΛΟ. Ευχαριστούμε. Και τώρα στον Μάρκ Ντίκ, μάνατζερ στο λιμένα του Ρότερνταμ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα. Το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και αποτελεί μεγάλο σημείο σύνδεσης με ένα πυλώνα προς την Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία, 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολούμε άμεσα 97.000 ανθρώπους. Ο σκοπό τη αρχή του λιμένα του Ρότερνταμ, για την οποία και δουλεύω είναι να βελτιώσουμε την η θέση του λιμένα του Ρότερνταμ ως κέντρο βιομηχανικής ανάπτυξης. Και λοιπόν επενδύουμε στην ανάπτυξη της χώρου του λιμένα για νέα ε, θέσεις ε, του λιμένα και για τις δημοσιοποδομέ και να περάσουμε τώρα στο TTIP. Στην παρούσα φάση 5,2% των ε, προϊόντων στους λιμένες μας έρχονται από τις ΕΙΠΑ ε, ως των ε, ανθράκας κοντέινερ και πετρέλαιο και περίπου 7,5% των προϊόντων που εξάγονται προς τις ΕΠΑ, προς που εξάγονται, εξάγονται προς τις ΕΙΠΑ. <coughs> Υπάρχει λοιπόν περιθώριο αύξησης του ποσοστού αυτού. Εν γέννη το λιμένα στο Ροτερντάμ αναμένει θετικέ ε, επιπτώσεις από την εφαρμογή του TTIP για την αρμόνιση των κανονισμών και η μείωση των δασμών θα αυξήσει το εμπόριο και προφανώς θα επωφεληθούν πιο πολύ τα εμπόρια τα container και αυτό ιδιαίτερα ε, θα ωφελήσει τα μεγαλύτερα πλοία. Κυρίως περιμένουμε μεγαλύτερη αύξηση στα, στα χίλιν αγροτικά προϊόντα, στα χημικά και στη μεταφορά μηχανημάτων. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσεις του TTIP της ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών και επειδή είναι σημαντική η μεταφορά για την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης, θα ήταν χρήσιμο να αναλύσουμε τον αντίκτυπο του TTIP στον τομέα μεταφορών. Περίπου 45% των προϊόντων που περνάνε από το λιμάνι του Ροταρντάμ είναι πετρέλαιο, άνθρακας. Και έτσι λοιπόν η TTIP μπορεί να ωφελήσει εάν συμπεριληφθεί μία παράγραφος για τις ενεργειακές στο TTIP. Ωστόσο, πρέπει να εξαιρεθούν τα προστατευτικά μέτρα, όπως γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο άνθρακα στις μεταφορές και στην παροχή ενέργειας και γι' αυτό λοιπόν προωθούμε υποδομές LNG, υγροποιημένου αερίου, βιομάζας, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το τι μπορεί να ωφελέσει προ την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε συμφωνία σε ό,τι αφορά τη χρήση υγροποιημένου αερίου. αερίου. Τέλος, ε, βλέπουμε ενδεχόμενα ωφέλη του TTIP στην ε, συνεργασία τη αλυσίδα παραγωγή παραγωγής. Αν ε, βελτιώσουμε τη διευκόλυνση του εμπορίου και τις Ε, επικοινωνία στην ανταλλαγή δεδομένων. Αυτό θα ωφελήσει και τι θαλάσσιε μεταφορέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγατε ότι είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι αποτέλεσμα θα έχει το TTIP στι εισαγωγέ, γιατί δεν υπάρχουν σχετικέ μελέτε. σω θα μπορούσατε να κάνετε σύγκριση με άλλε εμπορικέ συμφωνίε που ήδη έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε παρατηρήσει πραγματική αύξηση στι ε, εισαγωγέ, στι εξαγωγέ, υπάρχει πραγματικά ανταγωνιστικά κάποιο πλέον έκτημα, έχετε προσλάβει πιο πολλά άτομα. Υπάρχει ένα γνωστό ποσοστό αριθμητικό στοιχείο για το λιμένα του Ροτερνταμ. για το πετρέλαιο που εξαγάγεται στην Νότιο Κορέα. Έχει αυξηθεί πολύ. Έχουμε και δηληστήρια για το αργό πετρέλαιο το οποίο περνάει σε πολλές περιπτώσεις από το Ρότερνταμ. Βλέπουμε λοιπόν εκεί μια ελαφριά αύξηση. Ωστόσο το αργό πετρέλαιο περνάει κυρίως από τη Βορεια Θάλασσα στην Νότια Κορέα. Άρα ως λιμένα δεν μπορώ να πούμε ότι είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Ίσως θα πρέπει να σας δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες το λιμένα του Ρότερνταμ δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο αντικτύπος συγκεκριμένα, αλλά συνολικά ως λιμένας ε, που φυσικά ζούμε από τα προϊόντα που διαμετακοντίζονται και έχουμε ασφαλώ και έντονα βιομηχανικά κλάστερτ, ότι ασφαλώ όσο πιο ανοιχτέ είναι οι αγορέ, τόσο πιο μεγάλη τα φέλη για μα. Αυτό εν γέννη. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι βασικοί πελάτες ε, του λιμένα του Ροβερντάμ, οι μεταφορικέ εταιρείε, η εταιρεία, οι εταιρείε διοργάνωση μεταφορών θα ήθελαν να ζητήσουν μεγαλύτερη μελέτη δικτύπου για το θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη, λέει η συντονίστρια, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα για το λιμένα του Να είμαι ειλικρινής. Ας έχουμε λοιπόν να φανταστούμε θεωρητικά ότι καταργούνται όλοι οι φραγμοί μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Άρα μεγάλες εξαγωγέ ή εισαγωγές έχετε τις υποδομές να αντιμετωπίσετε μια τεράστια αύξηση και ιδιαίτερος το θέμα του LNG. Ευχαριστώ. Καταρχήν είστε πρόσδεκτοι. Ελάτε όποτε θέλετε να μας επισκεφτείτε. Ανοιχτή πρόσκληση. Τώρα, για την ικανότητα, το δυναμικό μπορεί να είναι πρόβλημα. Έχουμε κάποια προβλήματα χωρητικότητας ε, στα βότια. Μετά την κινέζικη πρωτοχρονιά είχαμε μια μείωση, όχι τόσο σημαντική βέβαια. Για τους σε αποβάθρες ε, έχουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τώρα υπάρχει μεγάλη φόρτος εργασιών. Αλλά δημιουργήσαμε το Mass 2 επέκταση δηλαδή των ε, ζωνών και προβλέπεται περαιτέρω επέκταση των ζωνών του λιμανιού για το μέλλον. Φυσικά δεν έχουμε άμεση ανταγωνισμό με, τις αμερικανικές, ε, με τα αμερικανικά λιμάνια, αλλά με το Αμβούργο και ένα άλλο ευρωπαϊκό λιμάνι έχουμε πολύ υγιή ανταγωνισμό. Ε, έτσι θα μπορέσουμε κάλλιστα να αντιμετωπίσουμε αύξηση, την, τη διαχείριση της αύξησης των, ε, της διακίνησης που θα προέλθει από το TTIP. Κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Δήμς, ε, Διευθυντής Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ε, σας παρουσιάσω εδώ τις απόψεις μας για τις μεταφορές και το περιβάλλον. Ε, είμαστε ένας οργανισμός που έχουμε την έδρα μας στις Βρυξέλλες και ασχολούμαστε με τις μεταφορές ε, και για να παρουσιάσουμε τις πραγματικές μας ενισχύσεις συμμετέχουμε και στις συνομιλίες TTIP. Για τη σημερινή εκδήλωση το τι μπορεί να κερδίσει η Ευρώπη από το TTIP είναι η ευκαιρία να έχουμε κάτι θετικό από όλα αυτά. Θα προσπαθήσω να τα καλύψω όλα σε πέντε λεπτά. Όπως έχει υποθεί στη συμβουλευτική ομάδα πάνω από ένα χρόνο τώρα, ε, ένα από τα βασικά συμπεράσματά μα είναι ότι ο κατάλογο των προτεραιοτήτων μα και αυτά που θέλουμε να αποσπάσουμε από του Αμερικανού, που οι Αμερικανοί μας θέλουν να αποσπάσουν από εμά είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτή πολύ από αυτόν που θέλουν εκείνοι από εμά. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το άνοιγμα τη αγορά. Οι, Αμερικανοί έχουν το Buy American. Εμεί δεν έχουμε Buy Europe. Ε, Europe. Ε, το ίδιο και με τι εξαγωγέ πετρελαίου και αερίου. Εκείνοι εξάγουν, εμεί όχι, όπω είπε ο προηγούμενο ομιλητή. Ε, και δεν ε, περιορίζουμε την υπηρεσία των λιμένων, των πλοίων ή των αερογραμμών, ούτε κατά διάνοια ω ΗΠΑ. Αυτά είναι λίγα παραδείγματα από τι μεταφορέ που γνωρίζω καλύτερα, αλλά είναι μεγαλύτερο το θέμα. Το Διεθνέ Εμπορικό Επιμελητήριο επιβεβαίωσε ε, στον δίκτυο των διεθνών τιμών και αληθεύει αυτό, ότι αυτό αληθεύει, ότι το άνοιγμα του εμπορίου στις ε, χώρες αυτές σε μέγιστη κλίμακα του 6 ε, φτάνει το 2,5 αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε το 2,2 πολύ χαμηλότερο και για να μεταφράσω τα αποτελέσματα είμαστε δύο φορές πιο ανοιχτοί ως προς την ε, πρόσβαση στην αγορά όπως θα έλεγε το Διεθνές Μελτιδιότητα ε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά γιατί απλώς δεν είμαστε Αμερικανοί. Καταλαβαίνω γιατί στην Ευρώπη πολλοί θέλουν ε, ίσω κανόνε παιχνιδιού, αλλά θέλουμε ίση αντιμετώπιση και από του Αμερικανού. Τι μπορούμε τώρα να αποσπάσουμε από αυτού. Ε, Σύντομε απαντήσει. Δεν έχουμε και πολλά να του δώσουμε σαν ταλλάγματα. Διότι αν δούμε τι δικέ μα περιορισμού στην αγορά, σχεδόν όλες, όλοι από του περιορισμού στην αγορά προκύπτουν από νόμου που ε, εφαρμόζουν πρότυπα διαδικασίε και υποδιαγραφέ ασχέτω από το που προέρχονται. Τα γενετικώ τροποποιημένα ε, λόγου χάρη δεν το επιτρέπουμε ούτε να το εισάγουμε από, την, από τους Αμερικανούς ούτε τα φέρνουμε. Το ίδιο και με το κρέας των χερμόνες ή με τα καλλιντικά ή με το πετρέλαιο που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Δεν μας αρέσει ε, να έχουμε τεράστια φορτηγά στους δρόμους μας που είναι πολύ επικίνδυνα για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τους ε, πεζούς και θέλουμε οι αερογραμμές να πληρώνουν το φόρο για τις εκπομπές διεξιδίου. Ε, στις Πολιτείες ε, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Είναι διαφορετικοί κανόνες μας για την πρόσβαση στις αγορές και δεν μας επιτρέπουν την πρόσβαση επειδή δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Ενώ εμείς δεν τους επιτρέπουμε λόγω των αρχών και των προτύπων μας. Οι γεωγραφικές μας ενδείξεις ήταν μια από τις λίγες εξαιρέσεις αυτόν τον κανόνα. Και πράγματι, αν ακούσατε τι λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε, τι λένε ότι θέλουν, επιβεβαιώνεται αυτό. Έχουν γίνει κάποιε ομιλίε για το TTIP και λένε ότι θέλουν περισσότερη επίδραση στις Αμερικα... από τι Αμερικανικέ εταιρείε στο πώ εμεί ετοιμάζουμε την νομοθεσία μα και να σταματήσει αυτή η πρωτοκαθεδρία των ευρωπαϊκών προτύπων με τους αρμόδιους ε, φορείς του ΟΗΕ όπου η Ευρώπη έχει ένα πολύ ε, μεγάλη βαρύτητα στην τοποθέτησή της. Ακριβώ επειδή τα πρότυπά τη επηρεάζουν. Ε, Εμεί λοιπόν θα θέλαμε οι Ηνωμένε Πολιτείε να μετακινηθούν από το 2,2 του ανοίγματο τη αγορά στο δικό μα 4,2 αλλά δεν είναι τόσο απλό, ε, δεν έχουμε τόσο πολλά να τους δώσουμε συνταλλάγματα εκτός από την υποβάθμιση των μα μας ε, προτύπων. Από τη δική μου λοιπόν τη σκοπιά η κίνδυνη η Ευρώπη να χάσει την αυτονομία της και οι φόβοι που υπάρχουν προ αυτό είναι κατανοητοί. Ε, έχουν Έχουμε πολλέ απαιτήσει για το άνοιγμα τη αγορά από την πλευρά μα, αλλά είναι λίγα τα ανταλλάγματα που έχουμε να δώσουμε. Ε, με το TFT να μην ξεχνάμε ότι οι καλύτερε συμφωνίε είναι αυτέ που ίσω δεν ε, πετυχαίνουν τον αρχικό σκοπό. Πώ θα μπορούσε το να ωφελήσει το περιβάλλον. Προφανώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να ευθυγραμμίσουμε το τι γίνεται εδώ και εκεί και να υπάρχουν αμοιβαία ωφέλη για το περιβάλλον. Να δώσω ένα-δύο παραδείγματα στον τομέα που γνωρίζω καλά, τι μεταφορέ. Ε, θα μ' άρεσε να υπήρχε ένα κεφάλαιο για την ενέργεια που να διευκολύνει τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την αποδοτικότητα. Όμω, εάν ε, διαπραγματευτούμε ένα τέτοιο κεφάλαιο, θα αφορά το να διευκολύνουμε τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το, τη βενζίνη και το, το αέριο. Θα ήθελα να υπάρχει μια διαδρατική συμφωνία για τις αεροπορικές εκπομπές ε, αέριου του θερμοκηπίου. Βλέπουμε να υπάρχει διάθεση για εμπορία, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει διάθεση αναχέτησης με κλιματικού στόχους. Γιατί να μην τους αναγκάσουμε να λάβουν την ευθύνη για τις μισές από τις διαστατικές εκπομπές. Ε, εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ Πολιτείες μας απαγορεύουν να έχουμε οποιοδήποτε περιορισμό στις εκπομπές εκτός τη επικράτειάς μα. Θα ήθελα οι Ηνωμένε Πολιτείε να ασχοληθούν με τι προδιαγραφέ για τα οχήματα σε διεθνέ επίπεδο. Όμω, όπως όταν δεν του βολεύουν, οι Αμερικανοί αρνούνται. Θα ήθελα επίση λιγότερε επιδοτήσει για τα ορυκτά καύσιμα ε, στι ΗΠΑ. Ε, και εμεί τα επιδοτούμε, αλλά πολύ λιγότερα. Εμεί σε κάποιε περιπτώσει θα πάμε χειρότερα από ό,τι αυτοί. Θα ήθελα και εμεί να έχουμε αμερικανική ομοσπονδιακή παρακολούθηση και έγκριση των οχημάτων. Ε, δηλαδή τα οχήματα να λειτουργούν ε, στο δρόμο όπως ε, στο εργαστήριο. Ή θα ήθελα προδιαγραφές για τις εκπομπές για τα οχήματα αυτά να είναι πιο αυστηρές όπως στην Καλιφόρνια. Είναι πολύ αυστηρότερες από τις δικές μας. Αλλά τα πράγματα αυτά δεν συζητώνται καν τα πλαίσια των συνομιλίων TTIP. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Το μόνο που συζητάτε εκεί είναι πώς να γίνει πιο περίπλοκο όταν φτάσουμε στου τόσους κανόνε, απαιτώντας και από τις δύο πλευρές να συμφωνούν ε, με παρα, παραλύοντας μέσω της ανάλυσης. Εδώ λοιπόν το TTIP είναι μια μεγαλύτερη προτεραιότητα από όλες τις ασιατικές μας συμφωνίες. Δεν είναι ούτε μέσα στο top 10 του Juncker τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Α, ανακεφαλαιώνοντας, ελπίζω να σας κατάλαβα ουσιαστικά όχι στο TTIP, έτσι δεν είναι. Είστε κατά το TTIP. Μακάρι να με πείσει κανείς ε, για το αντίθετο. Δηλαδή ότι η συμφωνία που θα καταλήξουμε θα είναι επωφελής για τους πολίτες και το περιβάλλον. Αλλά δεν έχω πει μέχρι τώρα για κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι όλες οι φιλόδοξες ε, προτάσεις δεν έκανε επιτάπητος. Ε, αποκλείονται από τις διαπραγματεύσεις σπάνια λέω όχι κατηγορηματικά για κάτι, ούτε και τώρα είμαι τόσο κατηγορηματικός, αλλά αν δείτε και το σχετισμό δυνάμεων, δεν βλέπω και πολλά ωφέλη για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα στο δεύτερο καταλογή που λέγατε τι θα ήθελα να δω μέσα στο DTIP, ουσιαστικά καταλήγατε σε πράγματα που είναι ανέφικτα. Τίποτα εφικτό βλέπετε, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για κάτι που θέλετε να συμπεριληφθεί στο DTIP και είναι και εφικτό ταυτόχρονα. Ίσως ε, το λιγότερο παρατροβηγμένο από αυτά που ζητώ, από αυτά που έχω στους καταλόγους μου, είναι να έχουμε παρόμοιες προδιαγραφές για τα οχήματα diesel τουλάχιστον, για τα αυτοκίνητα diesel. Μακάρι να έχουμε για τα αυτοκίνητα diesel τις ίδιες καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουν οι Αμερικανοί. Και να ανταποκρίνονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι με την πραγματικότητα. Έστω και μικρή πρόοδος είναι πολύ σημαντική. Άρα εσείς το τι το περιορίζετε στα αυτοκίνητα. Ε, θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτό που είπε πριν ο Μάρκ για, το, για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου α, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι την επιθυμία σας, τον πόθο σας για εναλλακτικέ πηγές ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από περιβαλλοντική άποψη όμως, ουσιαστικά είναι ένα καύσιμο ε, που έχει πολλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέψει να φτάσουμε στο στόχο του 2%. Στις ενεργειακές συζητήσεις υπάρχει ανισορροπία. Ουσιαστικά ευνοούνται τα ορυκτά καύσιμα γιατί τα περισσότερα καύσιμα περιέχουν άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα. Δυστυχώς η φόρο η ηλεκτρική ενέργεια ε, μένει εδώ, δεν μπορούμε να την ε, ε, έχουμε σε αντικείμενο εμπορίου. Και ακόμη και η βιοενέργεια περιλαμβάνει άνθρακα, ανθρακούχες εκπομπές. Οπότε δεν βλέπουμε την έκβαση των διαπραγματεύσεων να, ε, να εξυπηρετεί το στόχο της μείωσης των εκπομπών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το, ο μόνος υπέτης γι' αυτό είναι το εμπόριο. Το θέμα είναι ότι η, ορυκτή, η ενέργεια των ορυκτών καυσίμων είναι αντικείμενο εμπορίου, κάτι που δεν ισχύει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν, έχει, αν βάλουμε ενεργειακό κεφάλαιο στο TTIP, τι γίνεται με το αναπτυξιακό κεφάλαιο και το κεφάλαιο κυρίως αηφόρου ανάπτυξης. Θα έβρισκε σύμφωνο κάτι τέτοιο. Ναι, αν ε, ήταν απαιτητικέ ε, οι διατάξει, ναι, αλλά μέχρι στιγμή το θέμα τη εφόρου ανάπτυξη ε, δεν είναι και πολύ ρωμαλαίο στην TTIP. Ίσως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί, αλλά μάλλον απίθανο το βλέπω. Μάλιστα, τελευταίο τώρα λοιπόν. Τελευταία μάλλον, η κυρία Σαντρά Κρίνερ, η οποία είναι και αρχιτέκτονας και εργάζονται και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για το TTIP και την αρχιτεκτονική. Εγώ σπούδασα και στην Γερμανία και στη ΣΥΠΑ στο Πανεπιστήμιο της Κολόμπια και μετά επί σειρά ετών εργάστηκα σε διάφορε εταιρείε αρχιτεκτονικής στην Νέα Υόρκη, Πρωτού δημιουργήσω δική μου εταιρεία στην ΕΙΠΑ και εργάζομαι κυρίως σε εταιρικά project και εμπορικά project και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα που με αφορούν. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα ενδεικτικά της είπα ξεκινήσαμε το... στο Νέα Υόρκη την πρώτο κατάστημα Ισπανικής αλυσίδας ε, ενδυμάτων. Τα σχέδια τα έκανε Αμερικανός αρχιτέκτονας και εργαζόμουν για μια εταιρεία κατασκευαστική στην Νέα Υόρκη για το σύνολο της κατασκευής. Στη Γερμανία εκτελώ και ανοίγουμε καταστήματα αμερικανικής ε, αλυσίδας καφετέριας στη Γερμανία αλλά και στο Άμστερνταμ σε θετικές βάσεις. η τεχνογνωσία, η κατασκευή, τα σχέδια γίνονται από τη δική μου εταιρεία. Αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία ή την Ευρώπη. Στην Γερμανία υπάρχει μια ιεραρχία από τον αρχιτέκτονα, συμβούλους, σχεδιασμός, εκτέλεση. Στις ΗΠΑ υπάρχει διάκριση μεταξύ του σχεδίου και της κατασκευής. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μία εταιρεία στις ΕΠΑ που έχει πιο πολύ, είναι πιο πολύ υπεύθυνη για τις εγγύησεις. Στη Γερμανία υπεύθυνη από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου είναι οι αρχιτέκτονες. Νομίζω ο λόγος των οποίων στην παρούσα φάση υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στις πρακτικές μεταξύ ΙΠΑ και Γερμανίας είναι ότι οι Αμερικανοί Ήδη από την εκπαίδευσή του στις αρχιτεκτονικές σχολές ε, εστιάζονται πιο πολύ στην ιστορία, στην σχεδιασμό, ενώ οι γερμανικές σχολές εστιάζονται πιο πολύ στη δομική αρχιτεκτονική, όχι τόσο πολύ στις κατασκευές αυτές. Άρα, ένας ε, Αμερικανός τελειοφυτός, αυτό το αποφυτίσει μάλλον, έχει πάρα πολλά να μάθει και μόνο μετά από κάποια έτη μπορεί να ζητήσει άδεια αρχιτέκτονα, τις σχετικές εξετάσεις δηλαδή. Στη Γερμανία είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την πρακτική που περιλαμβάνει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και μπορούμε κατευθείαν να γίνουμε μέλη του αρχιτεκτονικού συλλόγου μετά από κάποια χρόνια άσκηση των κατοικών μας. Μπορούμε πολλά λοιπόν να μάθουμε ημένα από τους δε, από τα δύο διαφορετικά συστήματα και τις πρακτικές που ισχύουν στις δύο χώρες. Οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν πιο υψηλά πρότυπα εφαρμογής ανανεώσιμων ενεργειών. Έχουμε συγκεκριμένες γνώσεις αρχιτεκτονικής και επίπεδο αριστείας σε ό,τι αφορά τα δομικά υλικά. Οι αξιώσεις μας και οι προσδοκίες μας από τους πελάτες είναι επίσης διαφορετικές. για τα πιο υψηλά πρότυπα από τα οποία ισχύουν. Στη ΣΥΠΑ είναι πιο μεγάλη η αποδοχή, αν θέλετε, της πειραματικής αρχιτεκτονικής. Υπάρχει μια φιλοσοφική πτυχή και ανταλλαγή τέτοιων πειραματικών μορφών αρχιτεκτονικής. Αυτό γίνεται σεβαστό. Πιο ευρέως. Και είμαστε πιο αυθόρμητοι, πιο πρακτικοί στις λύσεις που αναζητάμε και είναι λιγότερο δεσμευτικοί οι κανόνες και οι κώδικες που μας ε, επιβάλλονται. Υπάρχουν και εκεί κάποια εμπόδια σε ό,τι αφορά το συνδυασμό κυρίως των δύο συστημάτων, των δύο υπήρων σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική. Ε, αλλά πιστεύω ότι είναι τόσο διαφορετική η εστίαση στα αρχιτεκτονικά ζητήματα στις δύο χώρες που θα μπορούσαμε αμοιβαία να επωφεληθούμε και οι δύο σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής φύσεως το οποίο τύφεται και σε επίπεδο δομικής ε, κατασκευής. Υπάρχουν λοιπόν τέλη και στη Γερμανία και στη ΣΥΠΑ, είναι διαφορετική διαδικασία διοδότησης ε, και η σχετική νομοθεσία, αλλά θα μπορούσαμε να εστιαστούμε στο μικρομεσαίο επίπεδο σε θέματα εκτέλησης για να ενισχύσουμε το επάγγελμά μας, την αναγνώριση των αρχιτεκτών παγκοσμίως μέσω των ανταλλαγών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, ένα από τα βασικά σημεία για τους αρχιτέκτονες, αλλά και για άλλους, για άλλα επαγγέλματα, θα είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Ώστε ένας Γερμανός αρχιτέκτονας θα μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπατε ότι οι Γερμανοί αρχιτέκτονες έχουν ε, Σπουδέ και μηχανικού ξέρουν να κατασκευάζουν, ενώ οι Αμερικανοί αρχιτέκτονε ασχολούνται περισσότερο με το design, με το σχεδιασμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με του Αμερικανού αρχιτέκτονε, αλλά δεν θα διάλεγα έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα για να μου χτίσει σπίτι. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή ε, στον τρόπο επικέντρωσης των σπουδών και στις, στις προτεραιότητες. Ε, στην, στις Ηνωμένες Πολιτι... Ε, στη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί σε θέματα μόνωσης, ε, ε, γνώσης μηχανικού, σε αυτά τα τεχνικά θέματα. Κάτι που δεν ισχύει στις Ηνωμένες δεν είναι τόσο απαιτητική. Και αν ζητήσετε από έναν αρχιτέκτο να σας κατασκευάσει ένα σπίτι, θα κάνει ένα καταπληκτικό σχέδιο, αλλά ακόμη και στην Αμερική θα προσλάβει έναν Ευρωπαίο αρχιτέκτονα για να εκτελέσει την κατασκευή. Και μάλιστα όταν ε, άνοιξα το γραφείο μου, ε, διαπίστωσα ότι ένας Αμερικανός αρχιτέκτονας ε, μπορεί να πάθει σοκ από το πόσες, πόσοι σύμβουλοι χρειάζονται και πόσα, πόσες πολεοδομικές άδειες επιμέρους. Στις ΗΠΑ έχουμε μία, ένα έντυπο στην, στη Γερμανία 15 πρέπει κάθε ο μηχανικός, ο, αρχιτεκτο, ο αρχιτέκτονας, ο μηχανικός ηλεκτρολόγος, ε, ε, κάθε ένας πρέπει να υποβάλει το δικό του σχέδιο για μονομένα τμήμα της πολυοδομικής άδεια. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική για τη Γερμανία. Πολύ πιο σημαντική ασφάλεια για τη Γερμανία από τι Ηνωμένε Αυτό είναι το συμπέρασμά σα. Όχι, εργάζομαι στη Γερμανία σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση και έχουμε πολύ πιο αυστηρούς κώδικες, ε, δηλαδή ε, αν ε, οι Αμερικανοί έχουν αυστηρότερες νομοθετικές διατάξεις, πρέπει αυτές να τηρούμε. Για φώτα, για παράδειγμα κάποιο φωτισμό εκτακτοναγκής ή, ή οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο απαιτητικέ. Έχουμε διπλάσιο αριθμό και απαιτήσεων στις Ηνωμένε Πολιτείε για το φωτισμό εκτακτών ανάγκης από ό,τι στη Γερμανία. Ναι, βέβαια, εσεί σπουδάσατε στι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι κάπω διαφορετικά, αλλά ένα Ευρωπαίο ε, αρχιτέκτονα που δεν έχει σπουδάσει στι Ηνωμένε Πολιτείε, τι βήματα θα πρέπει να ακολουθήσει τώρα, για παράδειγμα. Καταρχήν πρέπει να να ζητήσει πράσινη κάρτα. Μόνο με, έχοντας τέτοια πράσινη κάρτα μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει μέρος ε, σε εξετάσεις για να πάρει την άδεια. Και πρέπει πρώτα να έχει αποδείξει τριετή, ε, τετραετή πείρα απασχόληση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ίσως ε, με μια προσωρινή βίζα μπορεί να απασχοληθεί για ένα-δύο χρόνια και μετά να λάβει την πράσινη κάρτα και τότε μόνο μπορεί να υποβάλει την αίτηση για την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Και θα ακολουθήσουν 7 διαφορετικές εξετάσεις που είναι και δαπανηρές. Δυστυχώς το μικρόφωνο της ε, ομιλήτριας διακόπη ε, με υψηλό ποσοστό αποτυχίας και είναι διαφορετικές αναπολιτεία. Στην Νέα Υόρκη είναι πολύ διαφορετικέ οι εξετάσεις από ό,τι αντίστοιχες ε, στο Κεντάκι, στην Καλιφόρνια, στη Φλόριντα για τους αρχιτέκτονες για παράδειγμα. Από έγγραφα που κακώς ε, ε, διάβασα, δεν προκύπτει αμοιβαία αναγνώριση σε τέτοια επαγγέλματα όπως το, των αρχιτεκτόνων. Από τη στιγμή όμως που δεν θεά ε, εγκριθεί η αμοιβαία αναγνώριση. Ποιο θα είναι το δεύτερο καλύτερο βήμα. Συνεργασία. Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια. Από τη δική μου προσωπική επαγγελματική πείρα έχω μεγάλη περιέργεια για το πώς θα εφαρμοστεί το TTIP. Γιατί έχω συνεργασία με πολλά με πολλούς ε, εμπόρους ε, καταστηματάρχες στην Αμερική και θα ήθελα να ανοίξουν ε, καταστήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε ε, μεγαλύτερες ε, ευκαιρίες συνεργασίας με Αμερικανούς καταστηματάρχες στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Σας ευχαριστώ να κάλεσε τώρα τους βουλευτές να σχολιάσουν, να κάνουν ερωτήσεις και η συντονίστρια θα σημειώσει ποιοι ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο και στη συνέχεια θα κάνει μια σύνοψη. Η Αμα Μακλάκιν είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τη συντονίστρια, να ευχαριστήσω και τους ομιλητέ μας, τους σημερινούς. Νομίζω ότι συνολικά καταλαβαίνουμε από τις συζητήσεις ότι πολλά πιο πολλά μπορούμε να συζητάμε πέρα από το ISDS. Πάρα πολλές λεπτομέρειες υπάρχουν. Υπάρχει πραγματικά μεγάλο περιθώριο φιλοδοξίας, ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε θέματα αμοιβές αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να ωφελήσει πιο πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας τι ε, θέματα τηλεπικοινωνιών, ε, δημοσίων συμβάσεων και να απευθυνθώ ιδιαίτερα στον συνάδελφο από την Βιουρέκ, ε, ο οποίος δεν ήταν πιο σίγουρος για το ποια θα είναι τα ωφέλη και του καταναλωτές. Εγώ από τη δική μου πλευρά το να έχουμε μεγαλύτερη σε πιο πολλά προϊόντα, με πιο χαμηλό κόστος, με δημόσιες συμβάσεις που θα στοιχίζουν λιγότερο στο προλογούμενο και θα έχουν καλύτερους όρους, αυτό μου φαίνεται αρκετά αυτοπόδεικτο. Αναρωτιέμαι αν ο συνάδελφος έχει ήδη συνυπολογίσει τις ήδη φυστάμενες ε, συμφωνίες, για παράδειγμα με την Κορέα, ή αν έχει υπολογίσει συμφωνίες με τον Καναδά. Και βάσει αυτών των συμφωνιών μπορεί να εκτιμήσει το όφελος για τον καταναλωτή, γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι τα ωφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι η κίνδυνη. Ευχαριστώ πολύ, Βίκτορ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ απλώς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή την εκδήλωση. διότι εδώ και δύο ώρες κανείς δεν μίλησε για το χλωριωμένο κοτόπουλο. Δείχνουμε εδώ ότι ε, τα σοβαρά ζητήματα με την ε, πολύ γερή επιχειρηματολογία για το TTIP γενικώ και για το ISDS ειδικώ, καλώς τα θέτουμε, αλλά δεν έχουμε κάποιες λεπτομέρειες και έχω μια ερώτηση προς τους τρεις ομιλητές για την ε, κυρία από την Μισλά. Την ε, Σουηδή κυρία που εκπροσωπεί τα Σουηδικά Συνδικάτα και τον μάνατζερ από το Ρότερνταμ. Οι Σουηδοί και Ολλανδοί βουλευτές. Πού είναι όταν συζητάμε το TTIP και το SDS. Και με τους βουλευτές σας στις χώρες σας είχατε καθόλου συνομιλίες για να δείτε εάν γνωρίζουν τα προβλήματά σας και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας για να έχουν μια ορθολογιστική και σαφή και ακριβή απάντηση για τις γεωστρατηγικές μας ερωτήσεις, διότι το TTIP είναι γεωστρατηγικό ζήτημα της ε, ευρωατλαντικής μας οικογένειας, της Δύσης. Σας ευχαριστώ, Μπέρντ. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουν αρκετά... Επιφυλακτική όταν άκουσα για την ακρόαση αυτή. Αλλά είναι πολύ αναζωογονητική και δια... διαπιστώνω ότι αυτοί που πραγματικά δουλεύουν στον πραγματικό κόσμο έχουν άλλα προβλήματα, άλλες προτεραιότητες από ότι εμείς. Και γι' αυτό λοιπόν δεν θα κάνω οποιαδήποτε ερώτηση, αλλά θα κάνω μια διαπίστωση θα δηλώσω. Εσείς, από ό,τι φαίνεται, οι ομιλητές έχετε μεγάλη αποδοχή για το TTIP. Φυσικά με προτάσεις βελτίωσης. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Επιτρέψτε μου μία παρατηρήση. Δεν θα μιλήσω για τους ε, αρχιτέκτονες, αλλά είναι πολιτικός μηχανικός ο άντρας μου και εργάστηκε τέσσερα χρόνια στη ΣΥΠΑ. Έχει περάσει χρόνος βέβαια από τότε καιρός, αλλά έλαβε πράσινη κάρτα με δύο διπλώματα ε, πολιτικού μηχανικού. Βρήκε και εργοδότη γρήγορα, χωρίς να μιλάει τότε αγγλικά και ο εργοδότης του είπε «Δεν πειράζει, Μάικλ, κάτσε και να μάθεις ποια είναι τα πρότυπά μας. Και έμαθα ποια ήταν τα πρότυπα των είπα και ήταν πραγματικά πολύ ικανός, αν μεγάλη δεξιότητα σε θέματα στατικής, ε, για θέματα σεισμών. Και μετά από τέσσερα χρόνια με μεγάλη χαρά επέστρεψε στις είπα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ζαντού. Πρώτη παρατήρηση για τον Παρατήρηση για την ομιλία της κυρίας Μάστρομ που μας ε, είπε πάρα πολύ ωραία μας έβγαλε ένα κήρυγμα για το φιλελευθερισμό. 10% θα αυξηθεί η οικονομία τη Ευρωπαϊκή δεν θα υπάρχουν πια άνεργοι και το φιλελεύθερο μοντέλο θα συνεχίσει όπως είναι. Ωστόσο, το να χρησιμοποιήσουμε τον εκβιασμό της απασχόλησης για να λέμε στους ευρωβουλευτές ότι πρέπει να ε, αμφισβητήσουμε κάποια από τα στοιχεία της ε, διαπραγμάτευσης με τον Καναδά, αυτό το βρίσκω σκανδαλώδες και απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει πόσες θέσεις εργασίας παρήγαγε η συμφωνία με τον Καναδά και τότε να συζητήσουμε. Διότι αυτός ο εκβιασμός της απασχόλησης είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο. Ιδίως όταν ε, είμαστε εδώ για να προσπιστούμε το γενικό συμφέρον. Και δεύτερον, βλέπουμε πώς ε, διαμορφώνονται τα επιχειρήματα υπέρ της διατηρητικής συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα ήταν η απίστευτη ανάπτυξη. Η μελέτη, η πιο φιλόδοξη μελέτη που έγινε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 0,3% κέρδος ετησίως μελέτη που έγινε πρόσφατα και ελπίζω η εκπρόσωπο των Συνδικών Συνδικατών να την κοιτάξει αυτή τη μελέτη και να την διαβάσει πολύ προσεκτικά. Η μόνη μελέτη που βασίζεται σε όσα λένε και τα Ηνωμένα Έθνη για την απασχόληση στην Ευρώπη είναι κάτω από 6.000 θέσει εργασία και 223 θέσει εργασία θα χαθούν στι σκανδιναβικέ χώρε. Όταν γυρίσετε λοιπόν στη χώρα σα για να τα πείτε στου εργαζομένου σα, ελπίζω να του πείτε και αυτέ τι μελέτε και τα αποτελέσματά του. ίσω να εκπλαγείτε. Πάντω, εντυπωσιάστηκα που μα εξηγήσατε ότι υπάρχουν αυτοί που θα κερδίσουν και αυτοί που θα χάσουν. Για αυτού που θα χάσουν, τόσο το χειρότερο, ε, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση που θα πληρώσει τα σπασμένα. Εάν οι υπεύθυνοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων μιλάνε έτσι για την ιδιωτικοποίηση του, ε, της απώλειας και την ε, ε συλλογική ανάληψη του κόστους, αυτό το βρίσκω λίγο ε, απίστευτο. Τώρα, για τις προδιαγραφές και τα πρότυπα, δεν θα τι πειράξουμε λένε οι Ευρωπαίοι. Μα τι λέτε τώρα, τι διαπραγματευόμαστε αφού κανεί δεν θα πειράξει τίποτα. Ε, βλέπουμε ότι κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ πέρα. Εάν ε, όντω δεν τι πειράξουμε τι προδιαγραφέ και υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, ωραία. Ε, αλλά η οδηγία REACH αμφισβητείται κατά αυτόν τον τρόπο, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τι αμερικανικέ διαδικασίε για την αξιολόγηση του κινδύνου στι χημικέ ουσίε. Με τα χαρά να, να δεχτώ ότι ο όμιλο Μισλά, όπω και η υπόλοιπο βιομηχανία που ασχολείται με τα χημικά προϊόντα, χαίρομαι να δω ότι στηρίζονται το Ρίτ. Αλλά αλλά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αγωνιζόντουσαν για το ΡΙΤ, εσείς ήσασταν απέναντί μας. Τώρα μακάρι να έχετε περάσει στο τοπεδό μα, αλλά αυτή η αμοιβαία αναγνώριση νομίζω ότι σημαίνει ότι η προστασία τη υγεία θα πρέπει να ε, υπονομευτεί. Και όταν λέει η Ευρωπαία Επίτροπο δεν έχει κανένα επίπτωση στι νομοθεσίε μα, τρει εβδομάδε μετά τη σύναψη τη συμφωνία με τον Καναδά, τέλο πάντων ολοκλήρωσε την προσωρινή, μιλάω για την ε, συμφωνία με τον Καναδά, η Επιτροπή ε, ανέκαλε ανακάλεσε την ε, οδηγία για τα καύσιμα για να μην ε, ε, επιβάλλει πρόστιμα για τις ασφαλτούχους άμμους του Καναδά. Και στις Ηνωμένε Πολιτείες το ίδιο για τους διαταράκτες, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ενδοκρινικούς μάλλον διαταράκτες. Εδώ λοιπόν είναι πολύ μεγάλο διακύβευμα αυτό σήμερα, αλλά μην λέμε παραμύθια μεταξύ μας όταν έχουμε 27 εκατομμύρια ανέργους και κόσμο που υποφέρει και έναν ευρωπαϊκό λαό να ε, ικανοποιήσουμε. Κυρία Αρένα, ευχαριστώ. Όντως, Βίκτορ, δεν μιλήσαμε για τα χλωριωμένα κοτόπουλα α, στις ακροάσεις, αλλά ούτε για το ISDS μιλήσαμε. Οπότε οι καλεσμένοι δεν είπαν ότι το ISDS θα λύσει τα προβλήματα. Μην το ξεχνούμε και αυτό. Έχω μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο των Σουηδικών Συνδικάτων. Όντως, ε, μας είπατε ότι θα υπάρξουν νικημένοι και, νικητές και ιτημένοι. Το θέμα είναι να κάνουμε μια μελέτη επιπτώσεων ε, μετά τι διαπραγματεύσει, γιατί έγιναν μελέτε επιπτώσεων πριν τι διαπραγματεύσει, αλλά μελέτε επιπτώσεων για τι πράγμα. Δεν ξέρουμε το αντικείμενο, το, την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Το θέμα είναι να έχουμε μελέτε συνεπειών μετά τι διαπραγματεύσει, πριν την ψηφοφορία όμω. Για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε και μάλιστα όχι γενικέ ε, και αόριστες ε, μελέτες επιπτώσεων, αλλά μελέτες επιπτώσεων, τομέα, κλάδο, περιοχή, για να βοηθήσουμε τους ε, εργαζομένους που θα χάσουν ε, τις ε, θέσεις απασχόλησής τους. Στο Ταμείο Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίησης έχουμε 150, εκατομμύρια και δεν μπορούμε με αυτά να διορθώσουμε τα ολέθρια αποτελέσματα της αποκοσμιοποίησης. Ούτε μπορούμε να αυξήσουμε την προκοδότηση. Το Ταμείο όμως Προσαρμογής και Παγκοσμιοποίησης ενεργοποιείται όταν κάτι ήδη πάει στραβά. Δηλαδή ουσιαστικά βάζουμε ένα τσιρότο όπου μπορούμε όταν κάτι πάει στραβά. Αλλά η Σουηδική κυβέρνηση και τα Σουηδική συνδικάτα θα μπορούσαν να δεχτούν ε, με βάση την ανάλυση ε, κερδών ε, και ζημιών να δείξει μεγαλύτερη ελεγγύη προς τις χώρες που θα είναι οι χαμένοι από την όλη υπόθεση ώστε να τροφοδοτηθεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειοποίησης και να προλάβουμε τα προβλήματα, όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να τα επουλώνουμε όπως μπορούμε. Να πούμε από πριν ότι αν ένας τομέας πληγεί από την παγκοσμιοποίηση, να τον προετοιμάσουμε για μια εναλλακτική πορεία ή να, όπως προετοιμάζουμε τους εργάτες, ε, τους εργαζόμενους για ενδεχόμενο αναπροσανατολισμό επαγγελματικό. Γιατί λοιπόν ε, με τη λεγγύη να μην αντιμετωπίσουμε τα, αυτά τα προβλήματα. Είναι έτοιμα τα σουηδικά συνδικάτα να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους στον κλάδο που θα βγουν χαμένοι από το TTIP. Αν υποθέσουμε ότι αυτοί θα είναι οι κερδισμένοι. Ο κύριος Κρασνοντέμσκι. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Η ερώτησή μου απευθύνεται όχι μόνο στις ε, συναρπαστικές ε, παρουσιάσεις που ακούσαμε, αλλά ε, μία ερώτηση προς τους οργανωτές. Είχαμε πολλές ακροάσεις για το DTIP και διαπίστωσα ότι οι διοργανωτές δεν σκέφτηκαν να καλέσουν και από άλλες ε, περιοχές της Ευρώπης. Για παράδειγμα, ε, όπως δεν καλούσαν τις, ε, τους Πολωνούς πριν το 2004. Γιατί μιλήσαμε για το TTIP, για το σχέδιο του Γιούγκερ, το επενδυτικό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη έχει διευρυνθεί. Ε, γιατί δεν καλέσατε και καλεσμένου από τις ε, νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά νέες ναι, αυτές που μπήκαμε το 2004, γιατί και η Ρουμανία έχει αρχιτέκτονες και η Πολωνία, γιατί όλοι οι καλεσμένοι σας ήταν από τις ε, παλιές χώρες. Επίσης, το TTIP θα έχει διαφορετικές συνέπειες ε, για τις διάφορες περιοχές και χώρες της Ευρώπης. Οπότε, θέλουμε αναλύσεις και μελέτες για να δούμε πώς θα επηρεάσει το TTIP την κάθε χώρα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, την ε, πατρίδα μου, την Πολωνία, που είναι μια χώρα με μεγάλο πληθυσμό. Πώς θα την επηρεάσει το TTIP την Πολωνία. Μέχρι στιγμή δεν είχαμε πολλές εμπορικές συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο με ανατολικές χώρες είχαμε, με τη Ρωσία για παράδειγμα. Οπότε αυτό είναι το παράπονο μου και αυτή είναι η ερώτησή μου. Γιατί πώς τυχαίνει και σε τέτοιου είδους οργανώσεις, σε τέτοιου είδους ε, ακροάσεις δεν συμμετέχουν συνδικάτα από την Πολωνία για παράδειγμα ή εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων από την Πολωνία. Γιατί δεν με καλέσατε ε, εκπροσώπους επιχειρήσεων ή συνδικάτων από την Λετωνία για παράδειγμα. Thank you, thank you. Ε, κύριε Κέλλερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, τη συντονίστρια ένα, και σας ευχαριστώ που δοκιμάσαμε και κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες ακροάσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτά που ακούσαμε. Αλλά εξακολουθώ να αναρωτιέμαι τι ακριβώς θέλετε να μας φέρει το TTIP ως όφελος από Στη δική σας την πλευρά ακούσαμε τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και ακούσαμε ότι για παράδειγμα θα μας φέρει άρση των δασμών. Ότι θα εξοικονομήσουμε από τους δασμούς, θα το δαπανίσουμε και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απασχολήσουμε πιο πολλά άτομα ή θα δώσουμε πιο μεγάλους μισθούς, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, για τους εκπροσώπους του Λιμένα. Δεν άκουσα να έχετε μεγάλες προσδοκίες από το TTIP, πιο πολύ από το εμπόριο, αλλά όχι από το TTIP. Και πιστεύω ότι είναι μάλλον ε, προκαλεί σύγχυση το γεγονό ότι δεν είναι σαφές το τι μπορούμε να περιμένουμε από άποψη ανάπτυξης και μάλιστα Υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι δεν θα υπάρξει ούτε η ανάπτυξη, ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν σε ό,τι αφορά τις απασχόλησης. Θα χαθούν και δουλειές όμως. Μπορεί να μειωθούν και μισθοί. Και αυτό έχει αποτελέσει πόρισμα διαφόρων μελετών. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική απόδειξη των πλεονεκτημάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες και πολλά από τα μειονεκτήματα δεν έχουν καταρριφθεί. Σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, συμφωνώ για τα πιο υψηλά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, λέει ότι δεν θα πέσουν τα πρότυπα, θα αυξηθούν όμως. Εδώ δεν είναι σαφές ποια είναι η απάντηση. Για την ενέργεια Ξέρουμε ότι θέλουν μεγαλύτερη πρόσβαση, θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στα αρκετά καύσιμα στις είπα. και αυτό ισχύει. Αντίστροφος όμω, και οι αμερικανικές εταιρείε θα έχουν πρόσβαση στα δικά μα ορεικτά καύσιμα, τα οποία όμω εμεί ενδεχομένω δεν θέλουμε να τα κρατήσουμε σε πέταφος μα όπως για παράδειγμα θέματα υδρορογμάτευσης. Ίσως θα μπορούσατε να μου πείτε τι ακριβώς θα έχει ως όφελος νέες επενδύσεις, απασχόληση, μεγαλύτερους μισθούς, προστασία του κλίματος, προστασία του καταναλωτή. Πείτε μου και θα ήθελα με μεγάλη μου χαρά να ακούσω ποια θα είναι τα ωφέλη. Ευχαριστούμε. Από δική μου πλευρά, μία απάντηση για την κριτική ότι δεν είναι εδώ κανένα συνάδελφο από την Ανατολική Ευρώπη. Είναι τυχαίο. Είχαμε μία ακρόαση που διοργανώθηκε με την Επιτροπή Βιομηχανία, όπου ήταν εδώ δύο συνάδελφοι από ανατολικέ χώρε. Το θέμα δεν είναι να κοιτάξουμε τι ευαισθησίε των κρατών. Το θέμα είναι να βρούμε πού είναι το κοινό μα ευρωπαϊκό συμφέρον το συμφέρον των πολιτών. Να μην το το διάλογος αυτός. Ένα θέμα για τα πρότυπα. Θέλουμε αμοιβαία αναγνώριση. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό. Πώς θα αριθμίσουμε. Και πόσο μεγάλες θα πρέπει να είναι οι προσδοκίες κοιτώντα τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών σε διεθνεί επιτροπέ, σε ό,τι αφορά τα κοινά πρότυπα, δεν ε, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα πράγματα στις 14 Νοεμβρίου, Νοεμβρίου στην Γενέβη. Το UNCF ανέπτυξε νέα πρότυπα για τα ελαστικά το δέχτηκαν, τα δέχτηκαν τα πρότυπα αυτά σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη, εκτός από τη ΣΥΠΑ. Πόσο αισιόδοξοι λοιπόν μπορούμε να είμαστε για τη βελτίωση της κατάστασης από το TTIP. Και τώρα λοιπόν εσείς έχετε το καθήκον αγαπητή συντονίστρια να απευθύνετε τις ερωτήσεις αυτές προς τους ε, προσκεκλημένους. Ευχαριστώ. Δεν είναι απλό. Όταν κάποιο βουλευτή πριν το λόγο, δεν ξέρω αν έχει σχόλιο, ερώτηση ή ε, μείγμα. Έχω πολλέ ερωτήσει και σχόλια για τι μελέτε αντικτύπου. Και ακούστηκε και ιδέα μελέτη αντικτύπου. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαπραγματεύση τη συμφωνία, αλλά πρωτού κυρωθεί. Είναι κάτι που πιστεύετε θα μπορούσε να δουλέψει. Γιωχάνες, Εσένα ρωτώ, γιατί υπήρχε ένα συγκεκριμένο ερώτημα προ εσένα. Μπορεί να έχει κάνει τι δικέ σου μελέτε αντικτύπου για την συμφωνία με τον Καναδά. Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο. Υπάρχει μελέτη αντικτύπου για να δει αν είναι καλή για του καταναλωτέ. Νομίζω, εάν δείτε τον ε, προϋπολογισμό που χρειάζεται για να κάνει κανείς μελέτη αντικτύπου για μια συμφωνία σαν τη ΣΥΤΑ ή το TTIP ε, είναι πάνω από τις δυνατότητες μας, όχι δεν το έχουμε κάνει. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση της κ. Μακλάρκιν, να πω ότι προσπάθησα να εξηγήσω από προηγούμενες εμπειρίες μας ότι μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα, ότι ωφέλει από το TTIP θα υπάρξουν όπως οι τιμές, ο περιορισμός των δασμών, περισσότερη επιλογή, εμπορική διευκόλυνση και ούτω καθεξής. Αυτά μπορούν να ωφελήσουν τους καταναλωτές. Ελπίζω να το κατέστησα σαφές στο πρώτο πεντάλεπτο όπου τοποθετήθηκα. Αλλά αν δούμε τι ε, λένε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτήν την εμπορική συμφωνία, Μιλάμε για ένα μικρό τμήμα μόνο των διαπραγματεύσεων. Μιλάμε για τα, τα φρούτα στο δέντρο που μπορεί να πιάσει πιο εύκολα. Ε, καλό θα ήταν να ξεφορτωθούμε του τωρονιακού δασμού και βεβαίω θα είμαστε υπέρ αυτού του τρόπου διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, όμως το μεγάλο κομμάτι δουλειά για το TTIP είναι η μη δεσμολογική φραγμή. Εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με το οικονομικό κέρδος. Εκεί πρέπει να γίνει μελέτη αντικτύπου και να είναι και σαφή. Γιατί τα πράγματα δεν είναι σαφή. Οι ερευνητέ δεν ξέρουν καν πώ να τα καταμετρήσουν και να φανταστούν και θα είναι τα ωφέλη. Εάν δείτε λόγου χάρη τι εκθέσει τη Ευρω... Αμερικανική Επιτροπή, αυτό που ονομάζουν τεχνική φραγμή στο εμπόριο, αναφέρουν νομοθεσία, κανόνε, πρότυπα. Που δεν είναι απλώς τομείς όπου αν γίνουν ε, μικρές προσταφερέσει θα έχει κάνει καλύτερε τιμέ. Όχι, εδώ μιλάμε για πράγματα που είναι ουσιαστικά για την προστασία των ανθρώπων, των πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση της μείωση των δασμών και των τιμών που μπορεί να πέσουν ε, με ολόκληρο αυτό το πεδίο μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο. Ευχαριστώ. Η Σούζαν από τα Σουηδικά Συνδικάτα. Ε, και εγώ ξεπλάγει με τις δηλώσεις σου σήμερα και δέχτηκες και πολλά πειρά. Ε, όπως είπε και ο Γιάννικ, 600.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν ε, εξαιτίας του TTIP. Στη δική σου μελέτη υπάρχει τέτοιος αριθμός. Εσύ πώς το βλέπεις. Ο βουλευτής σας έθεσε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ξέρω ότι υπάρχει αυτή η πολύ αρνητική μελέτη για τις ε, επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και επίσης και για τις προοπτικές της αμερικανικής ανάπτυξης που είναι ανησυχητικότατη. Απ' την άλλη υπάρχει όμως και μελέτη πολύ θετική. Θα δημιουργηθούν πολλές θέσει εργασίας και για τις υπόλοιπες τρεις μελέτες την CPR και το ε, Εθνικό Επίπεδο επιμελητήριο της Σουηδίας και το CPR 2 εκεί οι μελέτες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα με διαφορετικά όρια. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί στις μελέτες, το δέχομαι. Όμως, καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν κάνει μια αποτίμηση των μελετών τη επιτροπή με τη σειρά του, όπου οι μελέτε τη Επιτροπή θα έπρεπε να θεωρούνται αξιόπιστε. Και εσείς είπατε ότι, α, εντάξει, είναι το καλύτερο σενάριο που, στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και μα δίνει μια μιακοπρόθεσμη, περιορισμένη, αλλά σαφή επίπτωση και άξιση τη ανάπτυξη που οδηγεί σε μακροχρόνια βελτίωση και στα θέματα ενεργείας. Ωστόσο, όταν συζητούμε με τους Αμερικανούς συνδικαλιστές για τις επιπτώσεις στην απασχόληση από τη Συμφωνία Ναύτα και το κατά πόσο η Συμφωνία Ναύτα επέτρεψε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Όταν λοιπόν αναλύουμε τις εμπορικές συμφωνίες, είναι πολύ νομίζω δύσκολο να απομονώνουμε μία σε σχέση με την γενικότερη διάθεση των εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε για θέσει εργασία, αλλά να δούμε αν είναι και ποιοτικέ. Τι είδου θέσει εργασία θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για να περάσει το θέμα τη καλή ποιοτική θέση εργασία. Όχι απλώ να υπάρχουν δουλειέ, Είμαστε πολύ επικριτικοί για την πολιτική λιτότητα και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ τα κάτι μελη Και μιλάμε για αλληλεγγύη με τον Νότο. Το έθεσε και άλλο μέλο του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό να αγωνιστούμε μαζί με του συντρόφου των συντηρητικών οργανώσεων για τι πολιτικέ τη Τρόικα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, καταστρέφουν το σύστημα συλλογικών συμβάσεων Μα το κάνουμε αυτό ε, και βεβαίω προεταθεί το θέμα. Αλλά το TTIP έχει πολύ δυναμικό και πρέπει να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να το εκμεταλλευτούμε. Να πούμε τώρα ναι ή όχι, να πούμε ναι, να δούμε τι μπορεί να μα προσφέρει το TTIP. Για όλους τους λόγους που ανέφερα, Εσείς τελικά θα αποφασίσετε αν θα πείτε ναι ή όχι. Και τελικώς η ερώτηση του κυρίου που μιλούσε για το χλωριωμένο κοτόπουλο. Έχουμε μιλήσει με τους Σουηδούς βουλευτές, αλλά θέλουν να μελετήσουν το θέμα περισσότερο. Την άνοιξη, την άνοιξη θα δούμε τι θα γίνει, είναι τότε κρίσιμα τα πράγματα και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους αρμόδιους βουλευτές μας. Ευχαριστώ. μία ερώτηση θα και προς εσάς ε, γιατί Μισλά και για τα ωφέλη που θα αποκομίσει από το DTIP. Και αυτό που εντυπωσιάζει και εκπλήσει μερικού είναι ότι αυτά τα κέρδη δεν θα επενδυθούν ε, ε, στην δημιουργία καλύτερων συνθήκων εργασίας ή στην αύξηση των μισθών. Μπορείτε να απαντήσετε. Βεβαίως για τον συνάδελφο που εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι δεν έχουμε εκπροσώπους από τις νέες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια μας βρίσκεται στην Πολωνία και έχουμε παρουσία και στη Ρουμανία. Και γι' αυτό η παρουσία μας είναι ευρεία. Είναι δύσκολο να δεσμευτούμε για μια συμφωνία που θα υπογραφεί που δεν ξέρουμε καν πότε αυτό που είναι σαφές είναι ότι επενδύουμε στην Ευρώπη και θέλουμε η Ευρώπη να, γίνει, να μείνει εξαγωγική βάση υψηλών προϊόντων, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και για να διαφυλάξουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα θα βοηθηθούμε από το TTIP. Θα είναι θετική η συμβολή του TTIP σε αυτό. Τώρα, αν αυτά τα κέρδη μεταφραστούν σε αύξηση θέσεων απασχόληση ή σε επενδύσεις, αυτό είναι δύσκολο ε, τόσο νωρίς να το προβλέψουμε. Γιατί οι συνέπειες συμφωνίας ε, θα αρχίσουν να φαίνονται μετά από μερικά χρόνια. Αλλά σίγουρα ε, θα είναι μια επενδυτική ενίσχυση η TTIP και θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει στο υψηλό επίπεδο εξαγωγών και τεχνολογίες. Είχατε επίσης επαφές ε, με ευρωβουλευτές. Προηγουμένως, ναι, βεβαίως, φυσικά με τους Γάλλους ευρωβουλευτές. Ε, τους εξήγησα αυτά που σας είπα σήμερα, ποιες είναι οι δραστηριότητές μας, τι κάνουμε σήμερα στη Γαλλία, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένε Πολιτείες και είχαμε και επαφές και με ε, Γερμανούς, ε, με Ρουμάνους, Ιταλούς, ευρωβουλευτές και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας. Πολύ ωραία. Τέθηκε και μία ερώτηση, μια στιγμή να ρωτήσει μου, στον εκπρόσωπο του λιμένα του Ρότερνταμ. Είπατε ότι δεν έχετε ε, ιδιαίτερες προσδοκίες από το TTIP, αλλά περισσότερο από την απελευθέρωση. Εννοείται ε, όσο περισσότερες εισαγωγές εξαγωγές έχετε, τόσο καλύτερα για σας. Ε, και αν αυτό επιφέρει συμφωνία, τόσο το καλύτερο. Όντως, ε, έχουμε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα και οι εισαγωγές εξαγωγές δεν περιορίζονται μόνο σε μια χώρα, είναι τεράστια γκάμα. Επίσης, 5% των συνολικών εξαγωγών και 7,5% των εισαγωγών είναι σχετικά χαμηλό τμήμα των εμπορικών συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι χαμηλές οι άμεσε εισαγωγέ και εξαγωγές και αυτό πιστεύουμε ότι με την που θα βελτιωθεί αυτό το ποσοστό. Φυσικά εμείς ε, είμαστε διευκολυντέ κατά κάποιο τρόπο. Οι επιχειρήσεις ε, που παράγουν τα προϊόντα στη Γερμανία και οι μεταφορεί που τα μεταφέρουν έρχονται στο Ρότερνταμ, εμεί απλώς εξασφαλίζουμε τη μετάβασή του στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι τόσο άμεση λοιπόν επιρροή μας. Απλώς διευκολύνουμε τις άλλες επιχειρήσεις για να φτάσουν τα επιχειρήματά του εκεί. Άκουσα κάποιες ε, παρατηρήσεις για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και ε, τα σχόλια του κ. Ντίξ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το λιμάνι του Ρότερνταμ επενδύει στι ε, υποδομές υγροποιημένο ε, φυσικό αερίο αλλά και στις εσωτερικές πλωτές οδούς γιατί είναι μια, ε, θέλουμε καθαρίες πηγές, ε, μορφές μεταφορών όχι μόνο από εσωτερικές πλωτές οδούς αλλά και ε, στις, στην ακτοπλοεία αλλά και τα μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης θα μπορούσαν να, να επενδύσουν ε, στις μεταφορές με υγροπημένο φυσικό αέριο γιατί είναι σχετικά περιβαλλοντικό, φιλοπεριβαλλοντικό καύσιμο. Βέβαια υπάρχουν οι περιορισμοί από το καμποτάζ. Γιατί για τα μεγάλα πλοία ε, δεν μπορούμε μόνο με ένα σταθμό να τα βγάλουμε πέρα. Και τώρα τα μεγαλύτερα πλοία με εμπορευματοκιβώτια έρχονται από τη Σιγκαπούρη. Πρόσφατα είχαμε το Όσκαρ 18.000 εμπορευματοκιβώτια σε ένα και μόνο πλοίο. Και 7.000 ε, ξεφόρτωσε στο Ρότερντα, μετά πήγε στο Αμβούργο. Αν θέλουμε καθαρότερες μεταφορές και διατλαντικά, η χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα πρέπει να διαβείται από πιο προστατευτικά μέτρα που θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια του TTIP. Αλλιώς τα πλοία δεν πρόκειται ε, που δεν είναι να επενδύσουν σε διατλαντικές μεταφορές με καθαρά καύσιμα. Ευχαριστώ και νομίζω ότι καλέσαμε λίγο πολύ όλες τις ερωτήσεις. Δεν ε, εξετάσαμε το πόσο αισιόδοξη θα έπρεπε να είμαι, αλλά αυτό θεωρώ ότι κύριε Λάγκα θα πρέπει να το αποφασίσει ο καθένα μόνο του. Σα ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάγκα για να α, ε, ολοκληρώσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλου του εκπροσώπου και τι εκπροσώπου ε, τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Ευρωπαίων Πολιτών σε σχέση με τι προσδοκίε που έχουμε για το TTIP. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντονίστρια. Ήταν πραγματικά χαρά μα που ήσασταν εδώ πέρα. Και νομίζω ότι έτσι δώσαμε ένα πιο ζωντανό χαρακτήρα στη συζήτηση από ό,τι στο παρελθόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τη γραμματεία για την προετοιμασία. Και θα τα, λέμε, θα τα πούμε λοιπόν αύριο το πρωί στι 9. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό σα βράδυ.